Bonjour, je vous remercie de prendre place. Καθίστε παρακαλώ. Σας καλωσορίζω για την πρώτη μας συνάντηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω να είστε όλοι σε καλή κατάσταση. Πριν ξεκινήσω με την ημερήσια διάταξη θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι τον καταστροφικό κυκλώνα ο οποίος χτύπησε την προηγούμενη νύχτα τα κράτη της Καραϊβικής, της Αντίλες και ιδιαίτερα δύο ευρωπαϊκά νησιά, το Σεμπαρτ και το Σεμαρτά. Το Σεμπαρτ και το Σεμαρτά έχουν καταστραφεί. Το Σεμαρτά έχει καταστραφεί κατά 95%. Το ίδιο ισχύει και για το Ολλανδικό κομμάτι και για το Γαλλικό κομμάτι. Δεκάδες χρόνια επενδύσεων στις χώρες αυτές έχουν ε, καταστραφεί πια. Αεροδρόμια, λιμάνια, υποδομές τηλεπικοινωνίας, τουριστικές υποδομές, όλα καταστράφηκαν. Και φυσικά υπάρχει και ο ανθρώπινος απολογισμός που δεν πάβει να είναι τραγικός. Και γι' αυτό λοιπόν είμαι βέβαιος ότι θα είστε όλοι αλληλέγγυοι μαζί μας και θα εκφράσουμε τα θερμά αλληλέγγυα αισθήματά μας προς αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και προς όλους τους λαούς της Καραϊβικής οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ξεφύγει από τις συνέπειες του δολοφονικού αυτού κυκλώνα, του Ήρμα και θα ζητήσω από τον πρόεδρο Γιούνκερ, την Επίτροπο Κρέτσου και ε, τον Επίτροπο Ντίμιτσα να κινητοποιήσουν όλα τα μέσα αλληλεγγύης προς τις χώρες αυτές. Ε, ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο γύρω από το ίδιο θέμα. Ο συνάδελφος Λαμπερτ Βανίστελ Ρόι. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε θα συμφωνήσω με αυτά. Εμείς συνεδριάζουμε στις Βρυξέλλες και βλέπουμε από μακριά τις συνέπειες αυτής της καταστροφής που προκάλεσε το Ήρμα. Και μάλιστα κινείται ο κυκλώνας προς τις Ηνωμένε Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς, τον, προς την γραμματεία. Ίσως θα μπορούσε να μας ενημερώσει σήμερα μια συνοπτική ανάλυση του τι έχει συμβεί στα διάφορα νησιά τα οποία ε, χτύπησε ο κυκλώνας, τι μέσα έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με αυτές τις περιοχές. Ε, δεν έχουν όλες οι χώρες αυτές τις ίδιες δυνατότητες ή τις δυνατότητες που απαιτούνται και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε Ευχαριστώ πολύ. Ζωζεφ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Εκπροσωπώ την εκλογική περιφέρεια αυτή που εφήγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι συγκινημένος από την συμπάθεια και την αλληλεγγύη η οποία εκφράστηκε προς τους πολίτες των περιοχών αυτών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Όπως είπα το Σέμαρτα έχει καταστραφεί κατά 95%. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Είχαμε ανέμους με ταχύτητα 300 χιλιόμετρων. Να σας θυμίσω ότι το 89 στα πλαίσια του κυκλώνα Χιούγκο ήταν ένα αεροπλάνο σταθμεσμένο στο αεροδρόμιο και με ανέμους 200 ε, χιλιόμετρων μετακίνησε το αεροπλάνο κατά 30 μέτρα, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται με 300 χιλιόμετρα. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε απτές αποδείξεις για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έτσι ώστε τα δύο αυτά νησιά που είναι δύο εξαιρετικά νησιά να μπορέσουν να, επιστρέψουν σε μια κάποια κανονικότητα και να μπορέσει ο κόσμος να επανέλθει σε μια κανονική ζωή. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει μια μικρή πρόταση για τροποποίηση και προτείνω και με τη συμφωνία των εισογητών της κυρίας Τζουφρίντα και του κυρίου Κοτσολίνο να αντιστρέψουμε τις εκθέσεις τους, να υπάρξει πρώτη η έκθεση Κοτσολίνο και μετά η Τζουφρέντα. Συνεπώς το 8 θα εξεταστεί πριν το 7 με λίγα λόγια Τώρα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 19ης ε, και 20ης ε, Ιουνίου, 29ης Ιουνίου, 12ης και 13ης Ιουλίου είναι διαθέσιμα online. Αν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θεωρούνται δεκτά. Επίσης μπορούμε να εγκρίνουμε το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής ΡΕΓΙ για το 2018. Η πρόταση έχει ήδη διανεμηθεί. Το να προγραμματίσει κανείς 20 συνεδριάσεις επιτροπών και υποεπιτροπών είναι δύσκολο και νομίζω ότι βρήκαμε τον καλύτερο τρόπο με ε, μία συνεδρίαση το μήνα εκτός ε, τον Αύγουστο και δεν υπάρχουν συνεδριάσεις την Πέμπτη το απόγευμα έτσι ώστε να μπορείτε να επιστρέφετε εγκαίρως στις εκλογικές σας περιφέρειες. Θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ψηφοφορίες λοιπόν για το 5, Γενικός Προϋπολογισμός, περίοδος Δημοσιονομική 2018. Έχετε όλη την κάρτα για την ψηφοφορία. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, εφόσον είστε έτοιμοι. Συμβιβαστική 1, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, η συμβιβαστική 1 γίνεται δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στο 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πέντε υπέρ κατά αποχές Προτείνω για τη συμβιβαστική υπαριθμών 5 να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. Περνάμε τώρα στην 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Λοιπόν επαναλαμβάνουμε. Α, για μια στιγμή. Διακόπτει ο πρόεδρος. Τροπολογία 20 λοιπόν τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Προτείνω ηλεκτρονικό έλεγχο για την 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθη με μεγάλη πλειοψηφία. Συνεχίζουμε τώρα με την 21. 21 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 26 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον για την 26. Ψηφίζεται. Τέλος. Μεγάλη πλειοψηφία. 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 34 ψηφίζεται. Τέλος. Adopté. Amendement 35. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 36. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Τελικά για την 36 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 37. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψήφος. Τέλος. Η έκθεση λοιπόν της Προέδρου μας ε, ε, γίνεται δεκτή. Συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία του συναδέλφου Βαλκαρσέλ. Δεν τον βλέπω. Δεν είναι παρόν αλλά έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσουμε αμέσως για να μην χάνουμε χρόνο. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 1. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. δεκτή. Παράγραφος 1, 1-10, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. AMC αγγλικά 2, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτό. Τοπολογία 3, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 33. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 52 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 58. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Προτείνω και εδώ ηλεκτρονική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 59. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική κλίση και επί της 59 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτή. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 77. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. Τελική ψήφος, ηλεκτρονική κλίση ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια στον συνάδελφο Βαρκάσελ. Bien. Notre collègue Geoffrida est, est arrivé, je la salue, et nous allons euh, passer à l'examen euh, de son... Λοιπόν, θα περάσουμε στην εξέταση της έκθεσης Τζουφρίντα, όπως έχει συμφωνηθεί για την ανταγωνιστικότητα στις περιοχές χαμηλού εισοδήματος και χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης. Θυμίζω ότι πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όπως γνωρίζετε όμως βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται με για τέτοιου είδους θέματα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν υπάρχει τρόπος βελτίωσης της πολιτικής συνοχής σε ορισμένες περιφέρειες της Ένωσης. Κάτι το οποίο θα έλεγα παίζει σημαντικό ρόλο για το σύνολο των πολιτικών των περιφερειακών. Όσοι συνάδελφοι δεν θα πάρουν μέρος στη συζήτηση, να φύγουν παρακαλώ, έτσι ώστε ο συνάδελφος να μπορέσει να παρουσιάσει ε, την έκθεσή του κάτω από ε, ανεκτές συνθήκες. Και μετά θα δώσουμε το λόγο στους σκιώδεις. Έχετε το λόγο. κυρία Τζουφρίδα. Λοιπόν, ε, για να ξεκινήσουμε, όπως είπατε, την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν και τα οποία σήμερα προσπαθούμε να καθορίσουμε σε λεπτομερέστερο επίπεδο, τουλάχιστον ως προς τις λεπτομέρειές τους. Η Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο για τις περιοχές που σημειώνουν, αν θέλετε, καθυστερήσεις και σε δύο υποσύνολα. Τα υποσύνολα αυτά περιλαμβάνουν τις περιφέρειες με ΑΕΠ που πλησιάζει τον μέσο όρο αλλά που δεν αυξάνεται πλέον και την περιφέρεια σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Και υπάρχει επίσης και μια διαφορετική κατηγορία χαμηλού ε, χαμηλής απόδοσης, ε, οι οποίες όμως ε, δείχνουν αυξητικές τάσεις. Είναι αρκετές οι περιφέρειες αυτές. Έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά η πολιτική την οποία ακολουθήσαμε μέχρι τώρα έχει αρχίσει να αποδίδει. Παραδείγματα. Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία κτλ. Η πρότασή μου καθορίζει κάποιους παράγοντες κλειδιά θα έλεγα που είναι αρκετά ευαίσθητοι και χρήζει να εξεταστούν και τις οποίες θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε. Το θέμα της εκπαίδευσης, το θέμα της κατάρτισης, το θέμα της απασχόλησης είναι θέματα τα οποία επανέρχονται και ξανά και ξανά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι η αναποτελεσματικότητα προκαλείται από τις αγορές εργασίας οι οποίες ε, είναι δίσκαμπτες εκεί όπου υπάρχουν και συλλογικές ε, συμβάσεις. Πιστεύει επίσης ότι και ο ελάχιστος μισθός, η ελάχιστη αμοιβή όπου είναι καθορισμένη δημιουργεί θέματα. Λέγει ότι δεν υπάρχει προοπτική ανάπτυξη αν οι επιχειρήσεις ε, δεν έχουν κίνητρα για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ο, θα έλεγα ο γόρδιος δεσμός εδώ είναι ο συντονισμός ανάμεσα στις εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές πολιτικές. Δεν έχω πολύ χρόνο και θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις σας πάνω στο ότι η Επιτροπή βασίζεται στη λογική της στο ότι το δημόσιο χρέος είναι το πραγματικό εμπόδιο στην ανάπτυξη. Η έκθεση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδέει το δημόσιο χρέος με το ρυθμό ανάπτυξης, λέγοντας ότι παρεμποδίζει τις δυνατότητες των περιφερειακών ταμείων να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι οι υποχρεώσεις ε, και οι δεσμεύσεις ε, που ε, δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβάλλει μειώνει τις δημόσιες επενδύσεις και οι περιοχές αυτές υποφέρουν κυρίως από έλλειψη επενδυτική. Αλλά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έλεγα ελείπουν ορισμένα στοιχεία και είναι τα θέματα που έχουν ε, σχέση με το έλλειμμα. Περισσότερο από το εθνικό δημόσιο χρέος, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί είναι σημαντικό θέμα και έτσι η πολιτική συνοχή δεν είναι σε θέση λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Τώρα, μακροοικονομικές συνθήκες. Δεν έχουμε χρόνο και δεν ξέρω αν θα ήταν απαραίτητο και χρήσιμο να διατρέξουμε την ιστορία μας πρόσφατα, αλλά η Ισπανία και η Πορτογαλία δείχνουν ότι είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε τη σχέση <clears throat> της πολιτικής συνοχής με τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί έτσι ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές που έχουν διαφορετικές δυσκολίες. Πρέπει να δούμε τις αιρεσιμότητες και στον τομέα της συνοχής και σε άλλους τομείς θα πρέπει να εξεταστούν έτσι ώστε να αριθμιστούν κάποιες ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν στο εσωτερικό της Ένωσης. Η ερεσιμότητα ισχύει και για άλλες πολιτικές, όχι μόνο για τις οικονομικές πολιτικές. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται όμως με θετικό τρόπο για να δίδει κίνητρα για μεταρρυθμίσεις. Και τελευταία τελευταίο κομμάτι ε, υπάρχουν ε, συσχετισμοί κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα στην πολιτική συνοχή από τη μία και τις ειδικέ αναχώρα εκθέσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να δημιουργούνται επιπλέον εμπόδια, ίσα ίσα θα έπρεπε να υποστηρίζονται μέσω του εξαμήνου περισσότερο οι περιοχές αυτές. Εκεί όπου η οικονομική ανάπτυξη είναι πάρα πολύ χαμηλή, οι συστάσεις θα πρέπει να είναι πολυετής και συμπεφωνημένες εκ των προτέρων με τις περιφέρειες στα πλαίσια μιας πραγματικής διαβούλευσης. Δεν θα πρέπει να μείνουμε στο να ορίζουμε κάποια σενάρια μετά την ανάγνωση της πρότασης της Επιτροπής. Βέβαια δύο εναλλακτικέ παρουσιάζονται. Από τη μία μια πολιτική συνοχής η οποία είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν επί τη βάση της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο βλέπει ότι η πολιτική συνοχής είναι κομμάτι και μέσο της οικονομικής ευρύτερα πολιτικής της Ένωσης. Το άλλο σενάριο λέει ότι η πολιτική συνοχή είναι προτεραιότητα για την Ένωση με διασφαλισμένη χρηματοδότηση και στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Οι επενδύσεις θα πρέπει να συμφωνούνται για τις περιοχές που παρουσιάζουν ειστέρηση και να διευκολύνουν την ισόρροπη και αηφόρο ανάπτυξή τους θα πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι έτσι ώστε να δώσουμε περισσότερες εγγυήσει για καλά αποτελέσματα μέσω θα έλεγα σχέσεων όχι υποταγής αλλά συνεργασίες των κοινωνικών πολιτικών με τις οικονομικές πολιτικές. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο θα ήθελα εγώ να προωθήσω. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τις παρενέσεις σας. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτό που μόλις υπόθηκε. Δεν υπάρχει συσχετισμός ξεκάθαρος και προφανής μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης και του επίπεδου ανάπτυξης. Μπορεί να υπάρχουν περιοχές που έχουν αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης, όμως ε, είναι ε, σε ιστέρηση ε, και δεν μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα υπάρχουν περιοχές με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που έχουν όμως ένα γενικότερο πλούτο ιδιαίτερα αυξημένο. Ο στόχος λοιπόν της πολιτικής συνοχής είναι ακριβώς να πάει προς την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δίνουμε τώρα λοιπόν το λόγο στο σκιώδη συγητή για το ΕΛΚ ο συνάδελφος, Φερνάντο Ρώσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την ε, πρωτοβουλία Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ελήφθη πριν από δύο χρόνια για πρώτη φορά με πιλωτικά προγράμματα στη Ρουμανία και στην Πολωνία, όπως ήδη υπόθηκε. Αυτά είναι σημαντική και πρακτική συμβολή σε μια πολιτική στρατηγική για αυτές τις περιφέρειες και την ανάπτυξή τους. Υπάρχει τώρα μια κατανομή σε δύο μεγάλες ε, ομάδες. Είναι οι περιφέρειες ε, με μια ε, μικρή ε, υστέρηση και οι περιοχές στο Νότο και την Ανατολή με μικρή ανάπτυξη. Τον Απρίλιο λοιπόν κατατέθηκε αυτή η πρόταση, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προτείνει μια μεγάλη ε, καινοτομία, είναι γενικά καλύπτει ευρύ φάσμα στοιχείων ε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές ώστε να αναπτυχθούν. Από την άλλη υπάρχει μια σειρά ε, περιοχών, μικρών αυτόνομων ε, περιοχών και δήμων που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κάθε περιφέρεια έχει τη δική της στρατηγική ανάπτυξης. Υπάρχουν λοιπόν ιδιαιτερότητες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι περιφέρειες να εμπλέκονται στις αποφάσεις. Όπως είπε και η συγγήτρια, οι ανθρώπινοι πόροι θα πρέπει να ενισχυθούν, να χρησιμοποιηθούν ε, και όλα αυτά μέσα σε ένα σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο. Άλλη μια παρατήρηση που έχω να, κάνει, να κάνω και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτό είναι ότι πρέπει οι πολιτικές ε, αποφάσεις να μας δίνουν καλύτερη πρόσβαση σε ε, ποιοτικά καλές πληροφορίες. Ε, αυτό το πράγμα το χρειαζόμαστε και το βλέπουμε ότι δεν είναι επαρκές και χαίρομαι που αναφέρεται στην έκθεση. Υπάρχουν περιοχές, για παράδειγμα η περιοχή στην οποία ζω, ε, όπου η ανάπτυξη είναι περιορισμένη. Ε, ο δήμαρχος ε, μπορεί να πρέπει να φροντίζει διάφορες τέτοιες περιοχές ταυτόχρονα. Και άλλες φορές υπάρχει και διαφορά μεταξύ των περιοχών που έχει στην αρμοδιότητά του. Είναι σημαντικό λοιπόν όλα αυτά, ε, το γεγονός ότι όλα αυτά αναφέρονται στο έγγραφο. Να αναφέρω και κάτι άλλο που το είπε η συνάδελφος. Στο δρόμο προς ε, την ε, σύγκληση υπάρχουν η αστική η ατζέντα για τις πόλεις και όλες αυτές οι πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να συντονιστούν για να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε περίπου ε, στη μέση της διαδρομής. Υπάρχουν ε, περιοχές ε, που βρίσκονται στο μέσο αυτής της διαδρομής και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την πραγματικότητα. Αλλά είναι ταυτόχρονα σημαντικό να είμαστε συγκεκριμένοι στις ε, πολιτικές μας για τις περιοχές ε, που έχουν αυτού του είδους τον πληθυσμό. Νομίζω λοιπόν ότι όλη αυτή η έκθεση καλύπτει όλα αυτά τα ιδιαίτερα προβλήματα, τα, τις πολιτικές, οικονομικές και διοικητικές ε, προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε και τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν ώστε να φτάσουμε στην σύγκληση και να έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία για την ε, λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων και εργαλείων και τη δημιουργία εργαλείων σε αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ ε, συνάδελφοι για τους ε, σοσιαλιστές. Κυρία Κράιλ, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω την εισηγήτρια σε όσα είπε. Υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ περιοχών με υστέρηση στην ανάπτυξή τους. Κατά τη συγγραφή της έκθεσης ήθελα να δω αν υπήρξε συζήτηση με την Κομισιόν σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε, σχετικά με τις περιοχές ε, οι οποίες οποίες έχουν πάρει πολλή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολλά χρόνια μέσα από τις περιφερειακές πολιτικές που υπάρχουν, αλλά δεν μπορέσανε να πραγματώσουν αυτή την ανάπτυξη. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να τους δώσουμε μια μικρή όθηση. Ε, για παράδειγμα, είχαμε πάει με την Επιτροπή μας στη Σικελία. Εδώ και δεκαετίες η Σικελία έχει υποστηριχθεί στεναρά όμως ξεκάθαρα βλέπουμε ότι δεν έχει καταφέρει να πάρει αυτή τη μικρή όθηση, το σπρόξιμο που θα την φέρει ε, μπροστά. Θα πρέπει ίσως να έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να θεσπίσουμε ώστε να υπάρχει πιο εντατική συνεργασία με τις περιφέρειες αυτές. Να οργανώσουμε κάτι το οποίο ε, θα ήταν μια συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξη για αυτές τις περιφέρειες. Ε, θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα ήθελα να δω αν μπορείτε να μας δώσετε μια τέτοια απάντηση μέσα από την έκθεση. Γιατί με ρωτάνε οι ψηφοφόροι μου ε, γιατί ε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλους ε, αυτούς τους ανθρώπους και να μην ακούμε αυτά τα χαζά επιχειρήματα των ανθρώπων που λένε να μην δώσουμε άλλα χρήματα πλέον. Καλό θα ήταν να μπορέσει η έκθεση να δώσει μια, ένα πιο ρεαλιστικό, μια πιο ρεαλιστική κατεύθυνση για το τι μπορούμε να πετύχουμε με την πολιτική συνοχής. Ευχαριστούμε. Για το ECR η κυρία Τόματσιτς δεν είναι εδώ. Για το ALDE ο συνάδελφος ε, Μπαργκέρ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το έγγραφο το οποίο υποστηρίζει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα τα οποία ακούω εδώ και πολλά χρόνια. Το βασικό μήνυμα είναι ότι χρειαζόμαστε πραγματική ανάπτυξη για να βελτιώσουμε τις στρατηγικές ε, ε, των περιφερειών. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η κυρία Κράιλ είπε ε, ότι πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει. Εγώ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε προγράμματα υποστήριξης της διαρθρωπικής μεταρρύθμισης. Ήδη πολλά χρήματα έχουν ε, δοθεί, ε, από ό,τι γνωρίζουμε από μια σχετική επιστολή για αυτά τα προγράμματα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω από την Κομισιόν ποια είναι η επένδυση που έχει γίνει, τι βελτιώσεις έχουν γίνει, γιατί αυτό είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτών των περιοχών. Τώρα, η μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, πολύ σημαντικό στοιχείο της έκθεσης. Νομίζω ότι έχουμε δει σε αυτή την Επιτροπή πόσο σημαντική είναι η μεταρρύθμιση στα εργασιακά. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, τη χώρα σας, προσπαθείτε να περάσετε μια τέτοια μεταρρύθμιση. Παρόλο που δεν υπάρχουν περιοχές σε υστέρηση ε, στην Γαλλία για μια χώρα με χαμηλά εισοδήματα. Τρίτον, αν ακούσει κανείς την εισηγήτρια καταλαβαίνει πως ναι μεν είναι ένα ε, έγγραφο εργασίας αυτό, όμως η μακροοικονομική, η πολιτική είναι αποφασιστική σημασίας για να έχουμε την απόδοση από τις επενδύσεις και η Κομισιόν σωστά λέει ότι πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση ε, με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τις πολιτικές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μακροοικονομικά. Και όπως επίσης και αν δεν κάνω λάθος, με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Κάνοντας ένα βήμα μπροστά μέσα από την ε, έκθεση αυτή, λοιπόν, θα μπορούσαμε να ε, συνδεθούμε με τα όσα ε, προτείνει η Κομισιόν. Αυτό το θέμα της μακροοικονομικής ερεσιμότητας είναι ένα θέμα υψής της σημασίας. Θα εμφανίζεται παντού. Δεν μπορούμε να, δίνουμε να κάνουμε επενδύσεις ελπίζοντας ότι απλώς κάτι θα αποφέρουν. Αυτό κάνουμε τώρα. Τελευταίο στοιχείο. Ε, θέλω να τονίσω κάτι που είπαν ε, και προηγούμενοι ομιλητές. Αν θέλουμε την ανάπτυξη αυτών των περιφερειών, θα πρέπει να δώσουμε μια έξυπνη εξειδίκευση. Πρέπει να επενδύσουμε σε περισσότερες δεξιότητες ανθρώπινες δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Εντάξει, να επενδύουμε σε υποδομές, αλλά μετά το 2020, με τα ταμεία συνοχής, θα έχουμε ήδη δώσει πολλά χρήματα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα που έχει δώσει η Κομισιόν σε αυτές τις περιοχές. Και ως καλός Ολλανδός να πω ότι οι αρχές στην, ε, στην κάθε χώρα θα πρέπει να, να αρχίσουν να βελτιώνουν τις διοικητικές τους ε, διαδικασίες ε, έτσι ώστε να παίξουν το σημαντικό ρόλο που έχουν να παίξουν σε αυτές τις περιοχές. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρη Παπαδημούλης. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τις περιοχές χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού εισοδήματο, Και υπάρχουν προφανείς ανάγκες να ενισχυθούν τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πόροι που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι εντυνόμενες ανισότητες. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τζουφρίντα διότι βάζει αυτή τη βάση στη συλλογική μας σκέψη. Και να υπενθυμίσω στον συνάδελφο από την Ολλανδία και τους φιλελεύθερους ότι ως καλός Ολλανδός πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα κονδύλια του EFSI είναι προτιμότερο να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που θα στηρίξουν την απασχόληση, το εισόδημα, την γενοτομία, την έρευνα στις περιοχές χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού εισοδήματος και όχι πανάκριβους αυτοκινητόδρομους όπως συμβαίνει στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εκεί πρέπει να πάνε τα λεφτά. Εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη θα σας δώσω έναν αριθμό, ένα στοιχείο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία που διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πηγαίνουν 78% στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, 11% στη νότια Ευρώπη και μόλις 1% στην ανατολική Ευρώπη. Και αυτό ενισχύει το brain drain στις χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης, αυξάνει τις ανισότητες, υπονομεύει τη δυνατότητα ανάπτυξης των περιοχών με χαμηλό εισόδημα και με χαμηλή ανάπτυξη. Και για να μιλάμε με ειλικρίνεια μεταξύ μας. Οι περιοχές χαμηλής ανάπτυξης βρίσκονται κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και οι περιοχές χαμηλού εισοδήματος στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία. Θα κάνουμε περισσότερα για να μειώσουμε τις ανισότητες. Θα ενισχύσουμε την πολιτική συνοχής. Ή απλώς θα λέμε σπαταλούμε εμείς οι πλούσιοι πολλά λεφτά σε αυτές τις περιοχές να δώσουμε λιγότερα. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να ενισχυθεί και να μην αποδυναμωθεί εν του νέου πολιετούς πλαισίου και ειδικά για αυτές τις περιοχές πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους και φυσικά να μην υπάρχουν σπατάλες και φυσικά τα, χρήματα να πηγαίνουν εκεί που θα πιάσουν τόπο και θα δημιουργήσουν απασχόληση αλλά γι' αυτό πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες που να ελέγχονται, αλλά και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία για να μπορέσουν αυτοί οι κανόνες να εφαρμόζονται λειτουργικά υποφελία της κοινωνίας. Και να δούμε και ορισμένα θέματα χωρίς τα χρωματιστά γυαλιά της σκοπιμότητας. Σε ποιο επίπεδο θα ορίσουμε τις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης. Να πω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, την Ελλάδα. Στην περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου Υπάρχουν τα νησιά της Ρόδου και της Κο που λόγω και του τουρισμού έχουν αξιοσημείωτα υψηλό εισόδημα σε σχέση με τους μέσους όρους και της χώρας μου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίδια περιφέρεια με νησιά που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, χαμηλή ανάπτυξη και έχουν ανάγκη αποστήριξη της δημιουργίας υποδομών. Θα καταδικάσουμε αυτά τα νησιά στη διατήρηση αυτής της χαμηλής ανάπτυξης και του χαμηλού εισοδήματος ή θα σκεφτούμε να ορίσουμε και σε χαμηλότερο επίπεδο από το ΝΑΤΣ 2 το πού ορίζουμε τις περιφέρειες χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού εισοδήματος. Και επίσης νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε ως Επιτροπή Περιφερειών ε, να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να δοθούν κίνητρα γι' αυτό και εργαλεία γι' αυτό ε, προς αυτές τις δύο κατηγορίες χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού εισοδήματο και από το EFSI και από το Horizon. Γιατί αλλιώς θα κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας και την ίδια ώρα θα αποδυναμώνονται οι πολιτικές περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Τζουφρίντα και να πω ότι εκ μέρους πολιτικής μου ομάδας ως κοιόδης εισηγητής επιδιώκω να συνεργαστώ με τους συναδέλφους όλων των πολιτικών ομάδων έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια καλή έκθεση που να στηρίζει αυτές τις περιφέρειες με την ευρύτερη δυνατή ε, συνένεση. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup, Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη. Το λόγο τώρα δίνουμε στους πράσινους, ο Γενής, συνάδελφός μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε μια ανταγωνιστικότητα παρόμοια σε όλες τις χώρες έτσι ώστε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην χαρακτηρίζεται από διαφορές μεταξύ των περιφερειών στο θέμα των εσόδων, για παράδειγμα. Όσον αφορά στο ΑΕΠ και την εσωτερική μετανάστευση που ε, δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι στην ουσία είναι μεγαλύτερο το κόστος όταν χτίζουμε νέες υποδομές ε, στις περιφέρειες όπου πηγαίνουν να εγκατασταθούν αυτοί οι εσωτερικοί μετανάστες, ε, αντί να τις δίνουμε τις επενδύσεις ε, στις περιοχές προέλευσής τους. Υπάρχουν 47 περιφέρειες σε 8 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στην ουσία έχουν χαμηλό επίπεδο ε, εισοδήματος και από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις, ε, οι περιοχές αυτές ε, αναπτύσσονται γρήγορα με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Απ' την άλλη, για να λυθούν τα προβλήματα αυτών των περιφερειών, η ίδια η Κομισόν ε, υπογραμμίζει στην έκθεσή της ότι πρέπει να γίνουν αυτά που μόλις ανέφερα. Νομίζω ότι οι περιφέρειες οι οποίες ε, δεν ε, αναπτύσσονται τόσο γρήγορα έχουν προβλήματα διοικητικά κατά κάποιο τρόπο ο τρόπος ε, στην ουσία που γίνεται, ο σχεδιασμός σε επίπεδο ευρωπαϊκό είναι αυτός που χωλαίνει. Θα πρέπει να φροντίσουμε όλες οι περιφέρειες ε, που βρίσκονται στις διάφορες ε, χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοιες ε, προκλήσεις, πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε τα αίτια αυτού του προβλήματος. Ε, αυτό το αναφέρει και η εκθέση της Κομισιόν. Είναι τα διάφορα κενά που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, για παράδειγμα. Νομίζω ότι αυτή η ανάλυση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να πετήσουμε λοιπόν από την Κομισιόν να κάνει μια πιο ενδελεχή και λεπτομερή εκτίμηση όλων των δυνατοτήτων που ε, έχουμε μπροστά μας ε, και να αναλύσει την εμπειρία μας. Θα πρέπει η Κομισιόν να έχει συνεχώς ε, πληροφορίες οι οποίες είναι ενημερωμένες. Ιδάλλως, οποιαδήποτε μορφή βοήθειας δοθεί, οποιαδήποτε μορφή αλλαγής γίνει στο νομοθετική βάση δεν θα έχει αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αίτια. Για κάποιες χώρες, ε, ας πούμε, θα χρειάζεται να έχουμε συγκεκριμένα, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Τέλος, να πω ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν αναφέρονται στο έγγραφο της Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να περιληφθούν στην έκθεση του Κοινοβουλίου. Είναι οι διαφορές σε επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών ε, του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά, μέσα στο ίδιο κράτος μέλος δηλαδή. Θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να αντικατοπτρίζονται στην έκθεση αυτές οι διαφορές. Ιδάλλως ε, δεν γίνεται να ζητάμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην ξεχάσουν αυτό το πρόβλημα, διότι φαίνεται ότι οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζονται ως ένα με την υπόλοιπη χώρα, παρόλο που υπάρχουν διαφορές σε σχέση με την γενικότερη κατάσταση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαματό για το FD. Η κυρία Ματώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Συζητάμε τώρα για περιοχές που υπολείπονται σε ανάπτυξη, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του Απριλίου που δίνει έμφαση σε 47 περιφέρειες σε αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που είτε έχουν χαμηλό εισόδημα είτε έχουν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. Βλέπουμε ότι οι περιοχές χαμηλού εισοδήματος είναι κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, ενώ οι περιοχές χαμηλού, χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης είναι κυρίως στο νότο. Η Επιτροπή λοιπόν αυτό που κάνει είναι να προσπαθήσει να δει με ποιο τρόπο θα ενισχύσει την περιφερειακή στρατηγική μέσω των διαφόρων ταμείων. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να βρούμε λύσεις. Συμφωνούμε ότι η Επιτροπή βρίσκει, θεωρεί ότι είναι πέντε λόγοι που ευθύνονται γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα οικονομική κρίση που έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία και έχει δημιουργήσει πάμπολες ανισότητες, ο χαμηλός ε, ρυθμός απασχόλησης, χαμηλός βαθμός ε, εκπαίδευσης των ε, κατοίκων, αλλά και ανικανότητα των θεσμών και της διοίκησης να ανταποκριθούν. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι στις χώρες αυτές, στις περιοχές αυτές δεν α, εκπαιδεύονται Τέλος, μια παρατήρηση πτώσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε αυτή τη λεγόμενη έξυπνη εξειδίκευση, ούτω ώστε να κλείσουμε το χάσμα μεταξύ των περιφερειών. Επενδύσεις λοιπόν στην εκπαίδευση είναι πολύ χρήσιμες, ούτω ώστε να καταστούν οι περιφέρειες αυτές πιο ελκυστικές να μπορέσουμε να αποφύγουμε το brain drain, αλλά η Επιτροπή κάνει ένα λάθος κατά τη γνώμη μου. Προσπαθούν να ενδυναμώσουν την πολιτική συνοχής Τα τελευταία τρία χρόνια όμως έχουμε επαναλάβει δεκάδες φορές τη συζήτηση αυτή. και όλοι καταλαβαίνουμε το ότι δεν υπάρχουν κυρώσει, ας πούμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ήταν ανάγκη να επιμείνουμε στο άρθρο 23. Έρχομαι... Ιταλία la pagina 18 del report, dove si descrive che nel solo periodo... έρχομαι λοιπόν από την Απολία και από το 2008 μέχρι το 2014 η μείωση των δημοσίων επενδύσεων στη χώρα μου έφτασε το 27%. 4% μείωση του ΑΕΠ, δύο επιπλέον σε σχέση με την υπόλοιπη Ιταλία, αν υποθέσουμε ότι το ΑΕΠ έχει νόημα πια. Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι όλες οι περιοχές και των 28 χωρών που παρουσιάζουν χρονική στέρηση βοηθήθηκαν από την πολιτική συνοχής. Ένα τμήμα των ευθυνών θα πρέπει να δοθεί, θα έλεγα, να απόδοθεί σε κάποιες πολιτικές κατηγορίες υπευθύνων που απέδειξαν επανειλημμένα την ανικανότητά τους αλλά θα πρέπει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να δούμε ότι επευλήθησαν κανόνες και για το ε, έλλειμμα και για το χρέος αντιπαραγωγική. Μείωση των επενδύσεων, το σημειώνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Γιατί να μην καταργούν πόδιο όδιο της συγχρηματοδότησης και γιατί να μην αφαιρείται το εθνικό κομμάτι της συγχρηματοδότησης από τον υπολογισμό του ε, ελλείμματος και του χρέους συνολικότερα. Λοιπόν, οι κοινότητες μας περιμένουν για την Ατζέντα 2020 τέτοιου είδους μέτρα, κίνητρα και όχι κυρώσεις. Και στο Μεντοτζόρνο, στη Νότια Ιταλία και σε άλλες περιοχές της Νότιας Ευρώπης πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις και συμπληρώσεις στην διοικητική τους μηχανή. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαφθορά μόνο μέσα από ένα ικανό προϋπολογισμό και με την επαρκή απλοποίηση θα υπάρξει μια συνεργασία ανάμεσα στις διαχειριστικές αρχές, τις πιστοποιητικές αρχές και τις εφαρμοστικές. Συνεπώς λοιπόν θα είμαστε στη διάθεσή σας ε, από εδώ και πέρα για το συγκεκριμένο ε, θέμα, τη συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι οκτώ έχουν ζητήσει το λόγο και μετά θα πρέπει να επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτριά μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε συνθετικοί παρακαλώ, σύντομοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώντας να ευχαριστήσω, λέει ο κ. Ζουλό την εισηγήτρια, η έκθεση της Επιτροπής είναι μια καλή έκθεση αν και πράγματι οι απόμακρες περιφέρειες ποτέ δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά στα πλαίσια των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό χρήζουν στήριξη οι προτάσεις. Δύο σημεία τα οποία κρίνω σημαντικά ανάμεσα και σε άλλα βέβαια. Πρώτον, η θέση η οποία δίδεται στην έννοια διαφοροποίησης. Είναι κάτι το αρκετά σημαντικό πρέπει στα πλαίσια της διαφοροποίησης να κάνουμε ε, βήματα. Πολλές φορές αναφερόμαστε στην περιπλοκότητα της πολιτικής συνοχής. Η περιπλοκότητα αυτή εν ολίγης οφείλεται στην ενιοποίηση των λογικών παρέμβασης και σε επίπεδο προγραμμάτων και σε επίπεδο περιφερειών ένα σημαντικό κομμάτι της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την διαφοροποίηση σε επίπεδο περιφερειών και όχι σε επίπεδο κρατών, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο εσωτερικό του κάθε κράτους μέλους υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις ανάμεσα στις περιφέρειες. Υπάρχει ας πούμε μεγάλη διαφορά στο Ile de France της Γαλλίας και την ίσο Μαγιώτου του Ινδικού. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε αυτά στα πλαίσια της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Ένα δεύτερο σημείο, πάρα πολύ συχνά γίνεται αναφορά στους λεγόμενους δείκτες της πολιτικής συνοχής. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη, δυναμικού τύπου ή μάλλον δυναμική στοιχεία και όχι μόνο στοιχεία στατιστικής. Πρέπει λοιπόν και τη διάσταση αυτή να μην την αγνοήσουμε. Και ένα τελευταίο σημείο είναι η σημασία η οποία αποδίδεται στην έκθεση για τη λήψη υπόψη των διαφορών. διαφορών. Νομίζω ότι και εδώ ε, είναι θέματα, βλέπουμε θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν για την προετοιμασία της περιφερειακής πολιτικής στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζουλό. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Καθώς οι περιφέρειες στην Βουλγαρία περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή, θέλω να συνεχίσω στην, να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, Πιστεύω ότι υπάρχει μια υποτίμηση του πόσο ειδικό είναι το πρόβλημα που υπάρχει σε αρκετές περιφέρειες της Ανατολικής Ευρώπης που υπολείπονται σε ανάπτυξη. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι περιφέρειες αυτές έχουν αποβιομηχανοποιηθεί σε ένα τεράστιο βαθμό. Στο παρελθόν υπήρξαν τεράστιες δομές, υπήρξαν επιχειρήσεις. Είχαμε ενεργό δράση στις εξαγωγές, υπήρχε χημική βιομηχανία, ο τομέας των τροφίμων ήταν ιδιαίτερα ανεργός και όλοι αυτοί οι τομείς έδιναν δουλειές σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Στην πορεία όμως μεταρρύθμισης του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος που ήταν ιδιαίτερα σημαντική μεταρρύθμιση, οι τομεί αυτοί κατέρευσαν, οι περιφέρειες αυτές κατέρευσαν. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο κείμενο για τη συνθήκη της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στο άρθρο 174, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική συνοχής θα πρέπει να επιλύει προβλήματα περιφερειών που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο. Πρέστιν με θερμινευόμενον ότι τα εργαλεία και τα μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν στις περιφέρειες αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Επομένως, ενίσταμε σε αυτήν την προσέγγιση που προτείνεται για περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για μακροοικονομικές στρατηγικές που θα φέρουν περισσότερες επενδύσεις. Όχι πως δεν χρειαζόμαστε επενδύσεις, όχι πως δεν χρειαζόμαστε τέτοια μέτρα. Δεν επαρκούν όμως αν δεν τα συνδυάσουμε με πιο στοχευμένες πολιτικές, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε νέες βιομηχανίες, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις βεβαίως. Θα βρεθούμε και πάλι απογοητευμένοι. Ο Επίτροπος Έτιγκερ στην παρουσίασή του, στις παρουσιάσεις του, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του α, φόρουμ για την συνοχή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, υπογράμμισε τα ακόλουθα. Προσπαθούσε να απαντήσει μια ερώτηση της συναδέλφου Κρέλ που ρώτησε πού πηγαίνουν τα χρήματα σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες αυτές. Και αυτό που είπε ήταν ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε, 60 cents από αυτό το ευρώ, επιστρέφουν είτε στη Γερμανία είτε σε άλλες α, βιομηχανίες των δυτικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μεθόδου εφαρμογής των μέσων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα τέτοιο επιχείρημα είναι καλό για την, κοινή γνώμη, για την αποδοχή της κοινή γνώμης στις δικές τους χώρες. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι να διαιωνίζεται η έλλειψη ανάπτυξης σε αυτές τις περιφέρειες που υπολείπονται. Οι πέντε λόγοι λοιπόν που προτείνει η Επιτροπή δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις πολύ ειδικέ συνθήκες. Προσωπικά λοιπόν είμαι υπέρ του να συνεχίσουμε να αναλύουμε, να συνεχίσουμε να εξετάζουμε πώς θα μπορέσουμε να υπερκάμψουμε αυτές τις ανισότητες. Και σημασίας μετά το 2020 η πολιτική συνοχής να είναι μια πολιτική δημόσιας επένδυσης. Επένδυση όμως που θα είναι στοχευμένη και θα συνδυάζεται με επενδύσεις βεβαίων ταμείων, ε, ιδιωτικών επενδύσεων, ιδιωτικών πρωτοβουλειών. Θα πρέπει να προωθήσουμε και να στηρίξουμε τις επενδύσεις αυτές μέσω ουσιαστικών στρατηγικών. Κλείνοντας, να σας πω ότι αν δεν ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό, τότε θα έχουμε να κάνουμε με επιπλέον εσωτερική μετανάστευση από την, εσωτερική, από την ε, Ανατολική με προς τη Δυτική Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ε, θέτουμε το ερώτημα γιατί μια περιοχή είναι ε, καθυστερημένη σε σχέση με την ανάπτυξη, υπάρχουν διάφορες απαντήσεις. Όμως, καλό θα είναι να μπορέσουμε να δούμε τις αιτίες. Όποιος ξέρει τις αιτίες μπορεί να λύσει και το πρόβλημα. Το Leibniz ε, Institute for Economic Research έκανε μία έρευνα και προσπάθησε ακριβώς να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα. Αυτό λοιπόν το Ίδρυμα, αυτό το Ινστιτούτο, βρήκε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν στην ιστέρηση της περιοχές. Αυτές οι περιοχές που λαμβάνουν ενίσχυση ε, μάλλον οι περιοχές που γυτνιάζουν με άλλες περιοχές που λαμβάνουν ενίσχυση ε, είναι λιγότερο ανταγωνιστικές και γι' αυτό έχουν υστέρηση στην ανάπτυξή τους. Αυτή η έλλειψη ανταγωνιστικότητας είναι που τις κάνει να υστερούν. Είναι εντυπωσιακό. Ε, θα έπρεπε η Κομισιόν να λάβει αυτό το αποτέλεσμα υπόψη της στην έκθεσή της. Εκεί που υπάρχει μεγάλη ε, ενίσχυση. Ε, στην ουσία ε, δημιουργούνται διαρθρωτικές και τεχνικές προκλήσεις για τους γείτονες. Είναι μια ανάλυση η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να μπει μέσα στο σκεπτικό μας. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την Κομισιόν αν γνωρίζει αυτή την έρευνα και να ρωτήσω και την συνάδελφο Τζοφρίτα εάν θέλει να τη στείλω αυτή την ε, έρευνα για να μπορέσει να διανθίσει περαιτέρω την έκθεσή της ε, βάσει αυτής. Νομίζω ότι έχει δίκιο το Ινστιτούτο. Και αν ε, έχει δίκιο, καλό θα ήταν να μπορέσουμε να βρούμε εργαλεία που θα μπορούσαν να στείλουν χρήματα σε αυτές τις περιφέρειες έτσι ώστε τα διαρθρωτικά ταμεία να δείξουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να προσθέσω και εγώ δύο-τρία σχόλια σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Στη συζήτηση αυτή, όταν μιλούσαμε για τις πολιτικές αυτής της περίοδου, ε, υπήρξαν διάφορες αμφιβολίες στο σώμα σχετικά με το κατά πόσο θα έπρεπε να δοθούν χρήματα σε αυτές τις περιφέρειες που τα σπαταλούν, ενώ υπάρχουν άλλες περιφέρειες οι οποίες είναι σε μεταβατικό στάδιο προς την σύγκληση. Αυτό ήταν το ερώτημα. Και καλό θα ήταν, αν θα θέλατε, να σας δώσω μια απάντηση. Ε, ίσως κάποιες ε, περιοχές να χρειάζονται πολιτικές που να είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους. Ε, χρειαζόμαστε όμως επιχειρήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτών των περιφερειών που δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Έχω λοιπόν μια πρόταση που είναι διτή. Πρώτον, έχουμε το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ε, οπότε μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε αυτό το πρόγραμμα και με μια περαιτέρω ενίσχυση ε, στα κράτη-μέλη μέσα από τεχνική βοήθεια, για παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι οι χώρες θα μπορούν αυτό να το χρησιμοποιήσουν. Ισπανία κτλ. Νομίζω ότι έχουν και αυτές αυτό το συμφέρον και ενδιαφέρον. Ίσως να είναι και ένα θετικό κίνητρο για να επενδύσουν και τα ίδια τα κράτη-μέλη, αν θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητες. Δεύτερον, γιατί να μην έχουμε ένα πιο προσγειωμένο εργαλείο. Οι περιφέρειες εθελοντικά να μπορούν να συνδέονται με μια άλλη περιφέρεια που δεν τα πάει τόσο καλά, για παράδειγμα, και με άλλες που τα πάνε καλά. Να έχουμε ένα τρίο, μια τριάδα περιφερειών που θα είναι δεμένες, συνδεδεμένες μεταξύ τους, θα μαθαίνουν η μία από την άλλη και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Στην Κίνα αυτό συμβαίνει υπάρχουν διάφορες περιφέρειες ε, που συνδέονται, αδελφοποιούνται ας πούμε με άλλες για να μπορέσουν να ανταλλάξουν εμπειρία. Δεν ξέρω τι έχει να πει η Κομισιόν γι' αυτό. γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε ένα καινούριο εργαλείο και αυτό το τρίο, η τριάδα των περιφερειών θα ήταν καλό, καλή λύση. Ο κύριος Παπαδάκης έχει το λόγο. Αλλά δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν νομίζω ότι το θέμα που βάζει η έκθεση επί της ουσίας και η παρουσίαση θέτει το ζήτημα της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη πρέπει να ρωτήσουμε για ποιον για τους εργαζόμενους, για το λαό ή για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί στη βάση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων δεν χωρούν υψηλά εισοδήματα. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας από μόνη της αναιρεί τον, τα υψηλά, δικαι, τα υψηλά μισθούς, τα εισοδήματα, τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Και απ' την άλλη, ε, Υπόθηκε εδώ το παράδειγμα των νησιών της ΚΟ και της Ρόδου ως παραδείγματα ανάπτυξης τέλο πάντων ενός αναπτυγμένα νησιά της Ελλάδας. Να θυμίσουμε ότι στην ΚΟ φέτος έγινε, έγινε σεισμός και με νεκρούς και με ε, σοβαρές υλικές ζημιές ε, σε ένα νησί που σφίζει από τουρισμό και ανάπτυξη έτσι όπως την εννοείτε εσείς και έτσι όπως χρηματοδοτείτε αφιδώς και την ίδια ώρα αντισυσμικά έργα δεν έχουν γίνει, είναι απαρχαιμένες οι υποδομές στο νησί ή στη Ρόδο, άλλο ένα παράδειγμα αναπτυγμένου τουρισμού, κερδοφορίας ομίλων και μια σειρά ε, ρεκόρ που γίνονται όλα τα τελευταία χρόνια, το 2013 είχαν γίνει πλημμύρες τεράστιες. Τα λέμε αυτά γιατί αντισυσμικά, αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι στην προτεραιότητα ε, των κονδυλίων, γιατί δεν αποφέρουν την κερδοφορία ε, που προσμένει το μεγάλο κεφάλαιο και ίσα ίσα δίνονται χρήματα και χρηματοδοτούνται κυρίως ε, επιχειρηματικοί όμιλοι ε, στη βάση ε, της λογικής των κερδών. Και νομίζουμε ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα και από ε, τα, την εισηγητική αναφορά που μίλησε για δισκαμψία επειδή υπάρχουν συλλογικέ συμβάσεις Άρα για δίσκαπτο ζήτημα είναι δηλαδή να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις σήμερα. Είναι δισκαμψία που πρέπει να αρθεί για να υπάρχουν κίνητρα για τους επιχειρηματίες. Βεβαίως αυτή η συζήτηση ε, είναι ε, σύμφωνη με τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεών της και στη Γαλλία που χτυπούν τώρα τις συλλογικές συμβάσεις ε, στις μαζικές απολύσεις, αλλά και στην Ελλάδα με τα αντεργατικά μέτρα που προωθεί συστηματικά όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση Ριζάνελ. Νομίζουμε ότι οι λαοί πρέπει να παλέψουν τα χρήματα που είναι ούτως ή άλλως δικά τους, να παλέψουν να γίνουν για τις δικές τους ανάγκες και όχι για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο Ζωζεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, πιστεύω ότι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε, θεωρώ ότι το είπατε ήδη αγαπητέ συνάδελφε, ποιες είναι οι αιτίε. Οι αιτίε μπορεί να είναι δομικές ή μπορεί να είναι α, συμπτωματικές υπάρχει η θέληση Είναι ανάγκη όμως να βρούμε ένα τρόπο να αντιδράσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε κατά νου αυτήν την πραγματικότητα για παράδειγμα, και των περιφερειακών χωρών που έχουν αρκετά μειονεκτήματα που προέρχονται από τη κλιματική αλλαγή, που μπορεί να είναι δομικά μειονεκτήματα. Η Επιτροπή θεωρώ ότι δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία όριζε πώς ακριβώς θα πρέπει να ασκηθεί η πολιτική συνοχής. σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Όλα αυτά καλώς τα έφυξε η Επιτροπή. Θεωρώ όμως ότι παράλληλα θα πρέπει η, Επιτροπή, η δική μας Επιτροπή να προτείνει κάποιες λύσεις που να είναι πιο σχετικές με τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν. Να μπορέσει να προτείνει και να εντοπίσει πιο συγκεκριμένες λύσεις, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις δυσκολίες της συγκεκριμένες των περιφερειών αυτών. Υπ' αυτήν την έννοια θέλω να συγχαρώ την συνάδελφο, την εισηγήτρια, η οποία έθιξε κάποια από αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε από κοινού για να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Ευχαριστούμε, το λόγο έχει ο συνάδελφος Έντμεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας άκουσα όλους ε, προσεκτικά και σκέφτηκα το εξής. Ο καθένας έχει δίκιο, είναι αλήθεια. Ε, θα πρέπει όμως να ξέρουμε πόσο συγκεκριμένοι, πόσο σίγουροι είμαστε για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για την ανάπτυξη των ε, περιοχών αυτών. Η λέξη κλειδί που ήδη υπόθηκε από προηγούμενους ομιλητές είναι οι περιφερειακές αρχές, οι τοπικές αρχές. Αυτές είναι που έχουν το κλειδί για την ανάπτυξη αυτών των περιφερειών σε υστέρηση. Πολύ συχνά σε τέτοιες ε, περιφέρειες και αυτό το ξέρουν όλοι και οι Κομισιόν και οι κεντρικές κυβερνήσεις. Ε, έχουμε το πρόβλημα με τις τοπικές αρχές. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ε, μοντέλο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτές τις περιοχές τις κάνει να πηγαίνουν προς τα πίσω. Ενώ ταυτόχρονα να βλέπουμε ότι στην ουσία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης σε τέτοιες περιφέρειες ε, που τις κάνει να εγκρίνουν πολιτικές και να τις ε, υιοθετούν παρόλο που δεν είναι πεπισμένες για την αποτελεσματικότητά τους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εμπιστευόμαστε περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι που πρέπει να φέρει την ευθύνη για όλα αυτά. Και στην συνέχεια μπορούμε να τις ε, κάνουμε να λογοδοτήσουν σχετικά με το αν έπραξαν σωστά ή όχι. Από την άλλη, αυτές οι τοπικές αυτοειδικήσεις μπορούν να καταλάβουν τις ε, εσωτερικές διαφορές εντός των ίδιων των χωρών. Στην Γαλλία, για παράδειγμα, άλλα μοντέλα έχουμε στο Παρίσι και άλλα στο νότο της Γαλλίας. Το ίδιο ισχύει και για την Πολωνία. Άλλα μοντέλα ανάπτυξη στη Δυτική, άλλα στην Ανατολική Πολωνία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη να δίνουμε περισσότερη ευθύνη στις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Δεν θα πρέπει να τις αναγκάσουμε να κάνουν αυτά που έχουν αποφασίσει κάποιοι άλλοι για αυτές. Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ρέγγιο. Έχει, αν έχουν αναφερθεί οι προλαλήσαντες στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούμε να σας δώσουμε το λόγο λοιπόν για να μας μεταφέρετε τις απόψεις σας. Thank you very much, Mr. President. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι όσο συντομότερο γίνεται αν και το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, να υπογραμμίσω καταρχάς ε, σαν ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η συζήτηση την οποία κάνουμε έχει υψηλό επίπεδο ευαισθησίας και περιπλοκότητας και είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσει κανείς όλα αυτά με απόλυτα ουδέτερο τρόπο. Από την άλλη εμείς δεν θέλουμε να ε, κρυφτούμε από τις δυσκολίες, να τις αγνοήσουμε και στον τομέα της πολιτικής συνοχής και στον τομέα της αναπτυξιακής γενικότερα πολιτικής της Ένωσης. Όπως υπογράμμισαν πολλά από τα μέλη της Επιτροπής σας, η έκθεσή μας υπογραμμίζει, σημειώνει τις διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες περιοχών, στην Ανατολική Ευρώπη και στον Νότο. Η επιλογή των ορίων και των κριτηρίων ήταν μια θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δύο κατηγορίες καλύπτονται πλήρως σε επίπεδο προτάσεων από πλευράς της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προετοιμάζουμε και μία επίσης ειδική ανακοίνωση για τις απόμακρες περιοχές, απότερες περιφέρειες Επίσης γίνονται πολύ και ενδιαφέροντα και στην Ανατολική Σλοβακία σε σχέση με περιοχές οι οποίες είναι ακόμα κάπως πίσω. Η στατιστική ανατολική πλευρά της Σλοβακίας έχει ξεφύγει αν θέλετε από την έκθεσή μας λόγω των συγκεκριμένων δικτών. Αλλά υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους εργάζεται η Σλοβακική κυβέρνηση με ενδιαφέροντα τρόπο. Αυτό που είναι σαφές λοιπόν εδώ είναι ότι οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ε, περιοχές αυτές ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της περιφερειακής απλά πολιτικής. Ε, θίγονται από τις οικονομικές γενικότερα εξελίξεις, από το μακροοικονομικό πλαίσιο, τις διαφροτικές μεταρρυθμίσεις και επίσης και την ποιότητα της διακυβέρνησης στην οικονομική δραστηριότητα οι επενδυτικές πολιτικές μπορεί να δώσουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα, τα αναμενόμενα συγγνώμη αποτελέσματα, εφόσον η διακυβέρνηση γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και θα συμφωνήσω με πολλούς από τους προλαλήσαντες ε, και αυτό μας δείχνουν τα ευρήματα, είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί κανείς με ένα μέγεθος για όλους, ένα νούμερο για όλους, αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν ισχύει και σε εθνικό επίπεδο. Ε, κάποιος από εσά είπε ότι ακόμα και στο εσωτερικό του περιφερειακού επίπεδου μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη και αρκετές διακυμάνσεις. Ε, αυτό το είδαμε και στα πιλωτικά προγράμματα με τα οποία δραστηριοποιηθήκαμε στην Πολωνία Εκεί στοχεύσαμε ε, το επίπεδο της πόλης, το επίπεδο του Δήμου, ε, για να μπορέσουμε να δούμε από κοντά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν ε, τη μία περιοχή και τη μία, τον ένα Δήμο από τον άλλο. Είδαμε λοιπόν το ότι να δαπανά κανείς χρήματα στα σωστά προγράμματα αυτού σαν δραστηριότητα δεν αρκεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπογραμμίσαμε τη μεγάλη σημασία να υπάρχουν οι συγκεκριμένες απαιτούμενες προϋποθέσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται τα συστηματικά θα έλεγα οργανικά εμπόδια που υπάρχουν και να αντιμετωπίζεται και το θέμα των προβλημάτων στην διακυβέρνηση σε ορισμένες περιοχές. Τον μήνα Οκτώβριο θα ε, παράγουμε το κατάλογο θα έλεγα ε, την ιεράρχηση της αξιολόγησης ε, της περιφερειακής διακυβέρνησης. Τώρα να επανέλθω σε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήσεις που τέθηκαν. Μία από αυτές είχε σχέση με μια έκθεση ενός think tank για τις επιπτώσεις στις περιοχές που υστερούν και την κατάσταση ε, την οποία αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις γειτονικές περιοχές που βρίσκονται σε άλλο επίπεδο. Εμείς εξετάσαμε την έκθεση αυτή. Ε, πρέπει να πω εδώ ότι έχουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο ε, τα οικονομικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν και κυρίως υπολογίστηκαν αλλά ακόμα περισσότερο θα πρέπει να πω ότι πάρα πολλές από τις πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν είχαν σχέση με την περίοδο 97-2007. Εμείς θεωρούμε ότι λόγω των βασικών διαφορών οι οποίες έχουν επισυμβεί από τότε, η έκθεση αυτή δεν ήταν όσο ενημερωμένη όσο οι προσπάθειες οι αντίστοιχες τις οποίες έχουμε κάνει εμείς πιο πρόσφατα. Ένα τελευταίο σημείο για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βανίστελ στον τομέα της συνεργασίας με τον οποίο θα συμφωνήσω φυσικά. Υπάρχουν πάρα πολλά και καλά παραδείγματα, ας πούμε η Ολλανδία, η Ρουμανία έχουν πολύ ενδιαφέροντα επίπεδα συνεργασίας. Θα πρέπει αυτά τα επίπεδα συνεργασίας να τα διευκολύνουμε έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται από κοινού και να μοιράζονται την εμπειρογνωμοσύνη την οποία κάθε περιφέρεια σωρεύει. Merci Σας ευχαριστώ πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ σύντομα να σχολιάσω κάποια θέματα. Να πω ότι η συζήτηση η οποία προηγήθηκε ήταν μια συζήτηση ιδιαίτερως πλούσια, η οποία καλύπτει όλα τα ερωτήματα και ε, αντιτίθεται μερικές φορές στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είδαμε επίσης ότι υπάρχουν μερικές φορές κάποιες αντιφατικές μεταξύ τους ε, αντιλήψεις στο εσωτερικό της πρότασης, αλλά αυτό το οποίο μετράει είναι να πετύχουμε τον βασικό στόχο που είναι η ανάπτυξη. Να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω στην συνάδελφο εισηγήτρια ότι τα κριτήρια και το ποσοστό ανάπτυξης ε, ε, αυτού δεν είναι ο στόχος. Δεν υπάρχει άλλωστε συσχετισμός προφανής τουλάχιστον ανάμεσα στον ρυθμό ανάπτυξης και στο επίπεδο ανάπτυξης. Στόχος και αυτοσκοπός δεν είναι ε, η ανάπτυξη αλλά είναι η απασχόληση. Εγώ προέρχομαι από την περιφέρεια της Ρεουνιό πριν από την κρίση του 2008 είχαμε ρυθμό ανάπτυξης 8% και όμως η χώρα μου πάντα ήταν πολύ πιο πίσω σε επίπεδο εξοπλισμού και υποδομών και το ίμιση του πληθυσμού της Ρεϊνιού ήταν κάτω από το επίπεδο έμβιας. Συνεπώς υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα στα οποία νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε και το οποίο δεν συζητιέται σήμερα είναι η χρησιμότητα της πολιτικής σύνοχης. Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία ανταπόκριση, απάντηση σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις και προβλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη για το σύνολο των περιοχών, όχι μόνο τις απότερες περιοχές, και θα είναι μια πρώτη βασική στρατηγική γραμμή η οποία θα χαρακτηρίσει το σύνολο της περιφερειακής πολιτικής. Και τέλος, δεν νομίζω ότι έχουμε επιμείνει επαρκώς εδώ τα προήμια στις προϋποθέσεις οι οποίες δεν τίθενται από πλευρά των κρατών μελών με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές να συνδυάσουν την δική τους επίδοση. Οι πολιτικές μας γίνονται μέσω παρεμβάσεων σε εδάφη τα οποία δεν είναι τα κατάλληλα προετοιμασμένα και συνεπώς οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται με την ευκολία που θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τζουφρίντα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ε, σύμφωνο πλήρως λοιπόν αυτά τα οποία μόλις είπατε Πρόεδρε. Το βασικό κλειδί ε, για να καταλάβουμε την κατάσταση και για να μην μείνει γράμμα νεκρό η προσπάθειά μας και για να μπορέσει η προσπάθειά μας να οδηγήσει σε ρεαλιστικές ε, καταστάσεις και μέτρα σε σχέση με τα προβλήματα είναι το να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα των διαφορών στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών εδαφών και στο εσωτερικό της πολιτικής συνοχής. Εσείς ε, απαντώντας και σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Κρέλ που δεν είμαι ανάμεσά μας τώρα, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική που θα πρέπει να βρίσκει λύσεις, λύσεις οι οποίες όμως να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα ερωτηματικά της κάθε περιοχής στα πλαίσια μια, ενός ευρυτέρου οράματος. Υπάρχουν περιοχές και στο νότο της Ευρώπης που παρά τις πολιτικές αυτές δεν μπορούν να καλύψουν την απόσταση που τους χωρίζει από το φορά Συνεπώς λοιπόν μέσω αυτή τη πρότασης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε και αυτό το κενό. Το κλειδί λοιπόν όπως είπα και ένα από τα σενάρια τα οποία έχουμε μπροστά μας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ερμηνεύσουμε την πρόταση της Επιτροπής είναι να υπάρχει υψηλότερο, ανώτερο επίπεδο διαβούλευσης με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι υπάρχει μια έντονη αντιστοίχηση ανάμεσα στις περιφερειακές πολιτικές και στις εθνικές πολιτικές. Να σας δώσω το ιταλικό παράδειγμα της χώρας μου. Στην Ιταλία δίδεται η μέγιστη δυνατή προσοχή, αναπτύχθηκαν στο παρελθόν συγκεκριμένες θεσμικές πρακτικές ε, για τις λεγόμενες συμφωνίες για την ανάπτυξη του Νότου, τα πάτη περιλσούντα. Ε, ε, πράγματι βοηθούν, συνεισφέρουν, στηρίζουν τις νότιες περιοχές της ε, Ιταλικής Δημοκρατίας όπου η οικονομική καθυστέρηση είναι μερικές φορές ενδυμική θα έλεγα. Επηρεάζονται θετικά λοιπόν οι περιοχές αυτές από τον σωστό προγραμματισμό σε εθνικό επίπεδο. Η ίδια λογική λοιπόν θα πρέπει να χαρακτηρίσει την ρουτίνα, την καθημερινότητα των δικών μας πολιτικών. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ομοιόμορφη απάντηση σε ετερόμορφες καταστάσεις. πως λοιπόν αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και από την συζήτηση η οποία προηγήθηκε ήταν μια χρησιμότατη συζήτηση, νομίζω δίδει πάρα πολλές φορές αφορμές για να γίνει η έκθεση όσο πιο αποτελεσματική γίνεται και έτσι θα προχωρήσουμε σε μια τελική πρόταση η οποία ελπίζω να τύχει της μέγιστης δυνατής πλειοψηφίας. Ευχαριστούμε. Να, να προσθέσω ότι η Επιτροπή μας έχει συμφωνήσει με την Επιτροπή Άγκρη για την εφαρμογή του άρθρου 53 του κανονισμού και η κυρία Τονισέλα η οποία δεν είναι σήμερα εδώ θα συμμετάσχει θα συμμετέχει στο εξή ε, σε κάθε συνεδρίαση η οποία ε, θα ασχολείται με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της συνεργασίας διάταξης. Η έκθεση ε, Αντρέα Κοτσολίνο που μιλά για τον ε, συντονισμό των μακροφεριακών, μακροπεριφερειακών πολιτικών. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Στα πλαίσια της προηγούμενης ε, συζήτησης υπόθηκαν πολλά. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα ήθελα να μιλήσω επί της ουσίας, θα ήθελα όμως να δώσω το περίγραμμα της δουλειάς την οποία κάνω. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν είναι ε, περιγραφική αν θέλετε ε, της, ε, του αντικειμένου όπως επίσης και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται οι συγκεκριμένες πραγματικότητες Να προσπαθήσουμε όμως, αυτός είναι ο βασικός στόχος, να βρούμε ένα πλαίσιο σταθερότερο για την εφαρμογή αυτών των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στο μέλλον. Και αυτά θα πρέπει να τα αποφασίσουμε τους επόμενους μήνες. Συνεπώς, Περισσότερο λοιπόν από μια έκθεση η οποία να έχει σαν βασικό στόχο την περιγραφή της κατάστασης είναι μια συλλογή των μεμονωμένων εμπειριών που έχουν μέχρι τώρα σωρεθεί και θα πρότεινα στους συναδέλφους ε, μια προσπάθεια επί τη βάση των στοιχείων τα οποία έχουμε ήδη για τρεις τομείς οι οποίοι κατά τη δική μου απόψη και εμπειρία έχουν σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά των μεμονωμένων περιπτώσεων και παραδειγμάτων. Τα τρία θέματα. Πρώτον, ας προσπαθήσουμε λοιπόν πρώτον να σχεδιάσουμε, να βρούμε μια πιο ισορροπημένη βάση διακυβέρνησης αυτής της στρατηγικής πώς θα μπορέσουμε εμείς να συσχετήσουμε τις βέλτιστες δυνατές πρακτικές που μπορεί να προέλθουν από τις εμπειρίες. Οι τρόποι που θα γίνει αυτό είναι διαφορετικοί. Πολλές φορές έχουμε την άμεση εμπλοκή των κρατών, άλλες φορές μόνο των τοπικών αρχών. Άλλοτε του ευρωπαϊκού επίπεδου σχεδόν άμεσα άλλο έχουμε παραδείγματα συνεργασίας του κράτους, της κρατικής μηχανής δηλαδή με τις περιφερειακές δομές. Από αυτή την πλευρά λοιπόν μπορούμε νομίζω να δούμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά, έναν μύτο ο οποίος θα μας οδηγήσει σε μια συνολικότερη αντίληψη της εμπειρίας για την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών. Ένα δεύτερο θέμα ε, κυρίαρχο είναι η συμμετοχή των κρατών μελών και σε σχέση με το ποσοτικό κομμάτι, το οικονομικό και σε σχέση όμως με το λεγόμενο ε, μακροοικονομικό πλαίσιο ή μάλλον χρηματοδοτικό πλαίσιο. Πώς μπορούν οι εμπειρίες αυτές να βοηθηθούν από ε, τους κρατικούς προϋπολογισμούς ουσιαστικά. Και τρίτον, το πλαίσιο των επενδύσεων τις οποίες έχουν ανάγκη οι μακροπεριφέρειες. Τι μπορούμε εμείς ε, να προσφέρουμε περισσότερο. Ε, από την εμπειρία που έχουμε τα τελευταία δέκα χρόνια, πέρα από τα μέτρα των διαφορετικών πολιτικών, τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε και μέσω των δημοσίων επενδύσεων και μέσω ελκυστικών για το ιδιωτικό κεφάλαιο επιχειρήσεων έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε όλο το δυναμικό το οποίο είναι διαθέσιμο για την ενίσχυση των πολιτικών αυτών. Ε, οι πολιτικές αυτές πέρα από τις δυσκολίες που συνάντησαν είχαν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα, προσέφεραν σε πολλές περιπτώσεις, αλλά αντιμετωπίζουν και ευαίσθητες δυσκολίες και καταστάσεις. Γι' αυτόν λοιπόν θα ακούσω με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις σας, θα κρατήσω από τις παρεμβάσεις σας και τις τροπολογίες φυσικά που θα καταθέσετε σε έφετο χρόνο, για να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε αν θέλετε κάποιες κατευθύνσεις για τις μελλοντικές πολιτικές για τις μακροπεριφέρειες. Τίποτα άλλο. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το είπες, αλλά η έκθεσή σου είναι στη συνέχεια της πρόσφατης έκθεση ε, ε, έκθεσης της Επιτροπής ε, 18 κράτη-μέλη και 3, 8 ε, τρίτες χώρες. Είναι λοιπόν μια μακροπεριφερειακή στρατηγική η οποία γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Δίνω τώρα το λόγο στο σκιώδη εισηγητή και μετά σε όλους όσοι θέλουν να παρέμβουν στη συζήτηση εκ μέρους του ΕΛΚ ο κύριος Μπόκοβιτς ο οποίος δεν είναι εδώ, άρα ο Λαμπέρτ. Ακριβώς αυτό που είπατε. Έχει σχέση με το έγγραφο. Ο Φρανκο Μπόγκοβιτς είναι στο Ιωταλίνε για το Προεδρείο Οπότε θα σας μιλήσω εγώ λίγο σχετικά με την περιοχή της Αδριατικής, για παράδειγμα, που είναι μια τέτοια μακροπεριφερειακή περιοχή. Αν δείτε την ιστορία της συνοχής, αυτή η εξέλιξη στη Βαλτική ξεκίνησε πρόσφατα και ακολούθησαν και άλλες περιοχές. Τώρα, το αν είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι, είναι παραπάνω από μισογεμάτο, γιατί αν δείτε τι έγινε στη Βαλτική, η οποία είναι μια ιδιαίτερα μολυσμένη θάλασσα, σε σχέση πάντοτε και με τη Ρωσία, και τι συνέβη μέσω αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων, ε, θα εντυπωσιαστείτε. Είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία σε πολλά επίπεδα ιδιοκτησίας βοηθά και στην Αδριατική. Υπήρχαν διάφορες συζητήσεις ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που αιωρούνταν έτσι. Ε, άμα δείτε τι γίνεται στην αλπική περιοχή, για παράδειγμα. Μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική βοηθά στην ανάπτυξη των μικρών χωριών. Μια πολιτική που έχει μεγαλύτερη σύνδεση. Αλλά αυτό που δεν κάνει και δεν πρέπει να κάνει είναι να στρεβλώνει την ευρωπαϊκή πολιτική γενικότερα. Δηλαδή ε, υπάρχουν κάποιοι που, θα, που πιστεύουν ότι αν πάμε σε μακροπεριφερειακό επίπεδο θα ξεχάσουμε τις απλές ε, περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Είναι μια προσέγγιση σε πολλά επίπεδα αυτή που θα πρέπει να ενισχύσουμε έτσι ώστε να ασχηροποιηθούν αυτά τα προγράμματα που αλλάζουν την κατάσταση πρώτα στις τυπικές περιφέρειες. Δεν είναι μια πολιτική η οποία ε, θα πρέπει να στρεβλώσει, να χαλάσει αυτά που ήδη έχουν συμβεί, θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. Τώρα, η στρατηγική επενδύσεων. υπάρχουν πράγματα που είναι καινούργια, όπως το ΕΦΣΥ. Όταν έχουμε τέτοια καινούργια πράγματα είναι πολύ δύσκολο να έρθουν στην επιφάνεια πρωτοβουλίες συνεργασίας ε, που να είναι τόσο στοχευμένη επένδυση που θα πηγαίνει στις δραστηριότητες των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Αν δείτε όμως τι γίνεται στη Βαλτική θα καταλάβετε ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο όσο πιο όριμοι είμαστε, τόσο πιο καλά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Όχι μόνο μέσω των ταμείων συνοχής, αλλά και μέσω των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η κυρία Μικελόβα ανεφέρθηκε στην Επιτροπή για την ε, ε, Εδαφική Συνοχή και πραγματικά πρόκειται για εδαφική συνεργασία. Ε, σύντομα τον Οκτώβριο θα έχουμε την 7η έκθεση για τη συνοχή που θα ορίσει την επόμενη περίοδο. Έχουμε λοιπόν την προσέγγιση αυτής της εδαφικής ε, συνεργασίας, την, περιφερειακή, ε, την εδαφική πολιτική και τις μακροπεριφέρειες. Όλα αυτά πρέπει να τα οριστικοποιήσουμε πριν ψηφίσουμε για την 7η έκθεση συνοχής. Και όπως είπε και ο συγητής προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πολιτική δέσμευση, να υπάρχει αίσθημα ιδιοκτησίας, να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνεργασία σε αυτούς τους τομείς και να ενισχύσουμε τη διοικητική ικανότητα των περιφερειών αυτών. Αυτό πάντοτε σε βάση απαρκών δικτών, για να μπορέσουμε πάντοτε να έχουμε μια βάση ε, τεκμήρια για τα όσα κάνουμε. Όχι άλλες μακροπεριφέρειες, απλώς ευάθυνση. Αυτό ε, λέω εγώ. Εντάξει, εγώ ως ε, Ολλανδός δεν θέλω τη Βαλτική, θέλω ξέρω εγώ τη Βόρεια Θάλασσα, γιατί είναι η δική μου θάλασσα. Δεν είναι αυτό τώρα να γίνεται. Καλό είναι να κάνουμε εμβάθυνση. Ευχαριστούμε πολύ τον Λαμπέρ. Για τους σοσιαλδημοκράτες, ο συνάδελφος Κλωσόφσκι έχει το λόγο. Πρόεδρε, εκ μέρους του κύριου Έμπα, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αναφορά. Αναγνωρίζω πραγματικά την σημασία αυτών των μακροοικονομικών στρατηγικών, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Η οικονομική κατάσταση σε πολλές από τις περιφέρειες έχει βελτιωθεί λόγω των στρατηγικών αυτών. Εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ενσωμάτωσης και είναι μέρος τη δέσμευσης, της δέσμευσης τοπικών και εθνικών αρχών εξίσου. Οι στρατηγικές αυτές όμως αντιμετωπίζουν και κάποιες προκλήσεις. Πρέπει, για παράδειγμα, να σκεφτούμε την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών συστημάτων που χρησιμοποιούμε. Και η αναφορά αυτή θα μπορούσε, η έκθεση αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως οδηγός για τη δημιουργία καινούριων μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη της Ένωσης, κράτη-μέλη, που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτού του τύπου τις ε, στρατηγικές. Πολλές φορές έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για συγκεκριμένες επαρχίες σε, επαρχίες που δεν, σε περιφέρειες που δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιου τύπου στρατηγικές. Τα θετικά σημεία της ε, έρευνας αυτής θα τα θίξουμε και στις ε, προτάσεις τροπολογιών. Ευχαριστούμε πολύ τον Σκιώδη. Ο Σκιώδης εισηγητής δεν είναι εδώ σήμερα γιατί άλλαξαν, άλλαξε λίγο το πρόγραμμα. Υπογραμμίζει όμως τη σημασία της έκθεσης αυτής, κυρίως ό,τι αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένων μακροπεριφερειακών στρατηγικών, αυτή της, αυτής της Ιωνίου θάλασσας για παράδειγμα. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική. Ένα δεύτερο συντομότατο σχόλιο, ο εισηγητής υπογραμμίζει το γεγονός ότι είναι ανάγκη να εμβαθύνουμε στην ανάλυση πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά τα μεταβατικά προγράμματα και πόσο στοχευμένα μπορούν να είναι. Υπάρχει ήδη χρηματοδότηση, κατά πόσο χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε στα χέρια μας αυτή την ανάλυση από την Επιτροπή, ούτω ώστε να δούμε με τι πόρους εφαρμόζονται οι στρατηγικές αυτές. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα, θα δούμε δηλαδή κατά πόσο λειτουργούν οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αυτές. Αυτά είναι βήματα που έχουμε ήδη κάνει στο Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι επαρκούν τόσο η χρηματοδότηση όσο και τα αποτελέσματα για την αριστερά έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστούμε το λόγο και ο κύριος Κοτσολίνο για τη δουλειά που έχει κάνει ε, μέχρι σήμερα. Ε, να πω ότι μας προσφέρει μια καλή βάση για να δουλέψουμε συλλογικά, γιατί όσα έχει επισημάνει και όσα συμπλήρωσε σήμερα δίνουν μια ε, σωστή, καλή, θετική βάση ε, για τη συνέχεια που πρέπει να δώσουμε με τη συμβολή όλων. Οι μακροπεριφέρειες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και είναι ανάγκη αν θέλουμε να συνεχιστεί με μεγαλύτερη επιτυχία να γίνει όλη η αναγκαία συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών εμπειρίας διότι τα αποτελέσματα είναι άνισα. Όπως υπόθηκε ήδη και από τον συνάδελφο Βανίτη στη Βαλτική έχουν προχωρήσει πολύ παραπάνω. Ε, άρα είναι χρήσιμο να δούμε πώς ε, στην περιφέρεια που με ενδιαφέρει περισσότερο που είναι η μακροπεριφέρεια Ιωνίου Αδριατικής μπορούμε να αντλήσουμε μια χρήσιμη εμπειρία. Επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από την πλευρά της ευρωπαϊκής στρατηγικής να μπορέσουμε, αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία που είναι και θετική και αρνητική, να διατυπώσουμε μια πρόταση για μια πιο συνεκτική και λειτουργική διακυβέρνηση αυτής της στρατηγικής. Ποιος κάνει τι. Job description δηλαδή. Πώς συνεργάζονται το ευρωπαϊκό επίπεδο, με το εθνικό επίπεδο, με το περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να έχουμε λειτουργικό αποτέλεσμα που να ανεβάζει την, ε, την απόδοση αυτής της στρατηγικής. Και εδώ έχουμε δύο σημαντικά πλεονεκτήματα δυνητικά αν αυτή η στρατηγική πετύχει. Γι' αυτό και πρέπει να επιμείνουμε στην ανάγκη να συνεχιστεί η, η στρατηγική των μακροπεριφερειών. Το πρώτο είναι ότι μας επιτρέπει να κάνουμε επενδύσεις που κάθε μια περιφέρεια μόνη της δεν μπορεί να κάνει ή κάθε κράτος μόνο του δεν μπορεί να κάνει. Πάρτε για παράδειγμα στην περιοχή Αδριατική Ιωνίου πόσο μπορεί μια επένδυση στις υποδομές, τις θαλάσσιες, να αναπτύξει τον τουρισμό ή την αλληλεία ή την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτές τις περιοχές επωφελία όλων. Και το δεύτερο α, κρυμμένο πλεονέκτημα είναι ότι αυτή η στρατηγική αφορά όχι μόνο κράτη-μέλη, αλλά και μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όμως έχουν στραμμένη την προσοχή τους, το ενδιαφέρον τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου και γειτονικά κράτη-μέλη που βρίσκονται, βρέχονται από την Αδριατική αλλά δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί έχει συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής να ενισχύσει τους δεσμούς με αυτούς τους λαούς, με αυτές τις χώρες, δείχνοντας ότι μέσα από αυτή την ανάπτυξη των στρατηγικών υπάρχουν προπές βελτίωσης της θέσης των πολιτών που ανήκουν σε περιφέρειες, κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα εργαλείο ε, εξαιρετικά χρήσιμο εκ μέρους της ε, Ευρωομάδας της Αριστεράς ε, έχω την πρόθεση να συνεργαστώ και με τον κύριο Κοτσολίνο και με τους ε, άλλους κοιόδη εισηγητές στη φάση της διατύπωση των τροπολογιών έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια έκθεση με την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία που να στηρίζει πάνω στη βάση των καλών πρακτικών και της ανταλλαγής εμπειριών αυτή τη στρατηγική. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ για τους πράσινους. Σκιώδης εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για μια εξαιρετική πρόταση. Εδώ και ένα χρόνο είχαμε ήδη εμείς κάνει μια έκθεση για την μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιουνίου και περιλαμβάνονται τα στοιχεία αυτά και στην σημερινή πρόταση. Ε, υπάρχουν ανησυχίες για διάφορα θέματα όπως η μεταναστευτική κρίση που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για αυτή τη μακροπεριφέρεια. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θέλω να σημειώσω για την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και τα ειδικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων περιοχών. Καταρχάς θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια λογική η οποία να έχει σαν στόχο τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το αίτημα να υπάρξει μια ενιαία κατά κάποιο τρόπο ευρωπαϊκή αντίληψη για το θέμα των μεταναστευτικών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ριζική πολιτική στο άσυλο, στην πολιτική του ασύλου, στην αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό εδώ να προασπίσουμε και την λεγόμενη blue economy. Η κιανή αυτή η οικονομία θα διευκολύνει εφόσον υποστηριχθεί σωστά και συνοδευτεί σωστά από δυνατότητες κατάρτισης που να λαμβάνει υπόψη της απαιτήσει συγκεκριμένων θέσεων, ε, κάποιες νέες δυνατότητες θα δημιουργηθούν, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές. Είναι απαραίτητο επίσης ε, να βελτιωθεί και το δίκτυο των διαθροτικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να είναι αηφόρος οικολογικά η παρέμβασή τους ανάμεσα στις περιοχές των χωρών που συμμετέχουν. Είναι επίσης σημαντικό σε όλες τις μακροπεριφέρειες να δούμε τι θα γίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς. Όπως είπαμε και πέρυσι οι στρατηγικές θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω της κινητοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων αλλά και των εθνικών δυνατοτήτων. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις διαφορετικές επενδύσεις, έχουμε το Ταμείο για την προενταξιακή βοήθεια μέχρι και το 2021. Υπάρχουν κάποιοι πόροι εκεί και πρέπει να γίνει σωστή χρήση. Άλλα χρήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι ο Horizon 2020 και το πρόγραμμα COSME. Σε επίπεδο διοικητικό όμως, τρικτό σένσο, να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω και τις προτεραιότητες που πρέπει να έχουμε. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τα εθνικά προγράμματα με τους στόχους της στρατηγικής. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Και τέλος, μια άλλη προτεραιότητα είναι η ανάγκη να εμπλέξουμε στη διαδικασία Αλήψεως αποφάσεων όχι μόνο τις τοπικές αρχές, τους δήμους, τις κοινότητες, έτσι ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον με συγκεκριμένες ρήτρες προστασίας, οδηγώντας τις περιοχές σε μια ευφυή, θα λέγαμε, μορφή ανάπτυξης. Ευχαριστώ, Χόβαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κοτσολίνο για την έκθεσή του. Η ανάπτυξη δικτύων σε διάφορα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε λιγότερο άτυπη βάση μπορεί να έχει μεγάλη αξία να φέρει πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω. Πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν σημαντικό ρόλο, θα προωθήσουν την συνεργασία, θα μας βοηθήσουν να μάθουμε από τις βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρία που έχουμε ως εκπρόσωποι των, του λαού σε πολλά επίπεδα και πολιτική να έχουμε δηλαδή μια περιφερειακή συνεργασία σε λιγότερο μακροεπίπεδο από ότι το Ηνωμένο Βασίλειο γενικά. Νομίζω ότι αυτές ε, οι στρατηγικές ε, έχουν διάφορες μορφές ε, με τις οποίες δρούν σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχει μια ευελιξία. Στη χώρα μου Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην ουσία είναι αυτή που διατάζει και ζητά όλοι να υποταχούν σε αυτόν τον τρόπο. Άρα η εναλλακτική αυτή είναι σημαντική για μας ε, και συμφωνώ πλήρως με τον συνάδελφο από την Ολλανδία. Γιατί βλέπω πόσο σημαντική είναι αυτές οι μακροστρατηγικές για τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών κρατών. Και εντάξει, έχει δίκιο λέγοντας ο συνάδελφος ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στη Βόρεια Θάλασσα, όμως μπορώ στο μέλλον να διαβλέψω κάποια προβλήματα τα οποία θα προκύψουν από το γεγονός ότι δεν θα είναι όλοι απαραίτητα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να κάνω φασαρία, απλώς έτσι θα γίνει. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν η Βρετανική κυβέρνηση είχε κάποιο όραμα, θα μιλούσε για μια συνεργασία στη Βόρεια Θάλασσα. Γιατί αυτό έχει σημασία όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για την Ιρλανδία που θα γίνει ακόμα πιο απομονωμένη στο μέλλον. Οπότε, μη μας, το μας ξεγράψετε ακόμα, γιατί στο μέλλον μπορεί να χρειαστούμε κάτι τέτοιο για να μπορέσουμε να έχουμε συνεργασία ταξί αυτών που είναι ε, πραγματικοί Ευρωπαίοι. Θα μπορούσαμε να, να ξεκινήσουμε μια ολόκληρη καινούργια συζήτηση βάσει της ε, εισήγησής σας. Από την DG Regio έχουμε τον Ζαμπιόν Άλκιν, τον καλωσορίζουμε. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια έκθεση για αυτές τις μακροπεριφερειακές πολιτικές. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεση. Έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα και με μεγάλη προσοχή ακούσαμε τα όσα είπαν ε, όλοι οι ομιλητές για αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να σας δώσω τώρα κάποια πολύ συγκεκριμένα δεδομένα που εξέφρασαν διάφοροι βουλευτές. Καταρχάς, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές ε, είναι μείζονος σημασία για τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Η στρατηγική για τη Βαλτιγική είναι από το 2009. Οι πιο πρόσφατες είναι αυτές για το Ιόνιο, την Αδριατική και την Αλπική περιοχή να σας ε, πω ότι στην ε, στρατηγική Ιωνίου Αδριατικής μόλις επιλέξαμε τα ε, project που θα χρηματοδοτηθούν. Εν τούτης, Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής που κατατέθηκε στις 16 Δεκεμβρίου και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, ε, υπήρξε ένα επιπλέον staff working document το οποίο παρουσιάζει κάποιες ποσοτικές πληροφορίες ε, σχετικά με την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών για να δούμε αν οι μακροπεριφέρειες ε, όντως κινητοποιούν ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια πέρα από την, και σε επίπεδο διεθνικής συνεργασίας. Σας δίνω το παράδειγμα της Βαλτικής που είναι το πιο προηγμένο. Όμως υπάρχουν διάφορα προγράμματα 60 έχουν ε, επιλεγεί. Τα 55 μας δείχνουν με ενεργό ε, τρόπο ε, να μας δείξουν ακριβώς πώς στην πράξη όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα. Το συνολικό ποσό είναι 3 300 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στα πλαίσια του πολυετού του δημοσιονομικού πλαισίου λοιπόν πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσπάθεια η οποία ως τώρα έχει φέρει σε εφαρμογή μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του προγράμματος. Υπάρχουν ε, πολλά σημάδια, βέβαια, ενθαρρυντικά για τις στρατηγικές αυτές. Ε, η ευθυγράμμιση μεταξύ της στρατηγικής και των πόρων της περιφερειακής πολιτικής που εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται μέσω των κρατών μελών απευθείας. Αυτά τα βλέπετε στην έκθεση της Κομισιόν. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ε, και να δίνουμε έναν απολογισμό των όσων επιτυγχάνουν αυτές οι στρατηγικές έτσι ώστε και σε δημοσιονομικό πλαίσιο να αντικατοπτρίζονται τα μαθήματα που παίρνουμε από αυτές. Να πω τώρα κάποια πράγματα σχετικά με κάποια ζητήματα που έχουν συζητηθεί πολύ. Είναι η διακυβέρνηση, η συμμετοχή των κρατών μελών και οι επενδύσεις και η σχέση τους με τις άλλες πολιτικές. Θα ξεκινήσω με το τρίτο στοιχείο με αφετηρία το γεγονός ότι οι στρατηγικές αυτές εξ αρχής ήταν θύματα των ανησυχιών που πηγαίνουν πέρα από τις περιφερειακές πολιτικές. Ας πούμε, στη Βαλτική ήταν ε, το περιβάλλον που γέννησε τη στρατηγική και έχουμε ήδη τα αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν μια, ε, μια διάσταση εγκάρσια των στρατηγικών που είναι πολύ σημαντική. Στο μέλλον υπάρχει σύσταση οι στρατηγικές να είναι πιο καλά αγκιστρωμένες στις ευρωπαϊκές πολιτικές π.χ. του περιβάλλοντος ή τη θαλάσσια πολιτική. Ε, η ενέργεια και οι μεταφορές είναι επίσης ε, θεματολογίες στην καρδιά των στρατηγικών, έτσι ώστε τελικά να υπάρχει ουσία ε, και στα αποτελέσματα και στο εύρος των στρατηγικών. Η Επιτροπή θέλει να ε, εκφραστεί για αυτό το θέμα. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να γίνει ίδια συζήτηση και για τις άλλες πολιτικές που είναι ήδη στη στρατηγική μας, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές. ή αν ε, θα έπρεπε γενικότερα να υπάρχει μια εγκάρση οπτική που θα μιλήσει ακριβώς ε, για για το εύρος και το πεδίο αυτών των πολιτικών. Τώρα για τη διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η διακυβέρνηση σε αυτές τις στρατηγικές. Ως τώρα είδαμε πως υπήρξε μια προσαρμογή Ε, ξεκίνησε η στρατηγική με βάση μια πολιτική συνένεση για την εφαρμογή, όμως οι, οι δράστες, οι, τα μέλη αυτής της πολιτικής ε, ήταν πολύ πιο εκτεταμένοι. Είχαμε μεν το κράτος, αλλά είχαμε και την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση ή όχι και ακούμε και τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σε αυτό. Κάτι άλλο ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη των πολιτικών είναι η συμμετοχή με ίδια κεφάλαια των κρατών μελών. Οι στρατηγικές είναι bottom-up, δηλαδή πηγαίνουν από κάτω προς τα πάνω. Θα πρέπει λοιπόν για να σεβαστούμε αυτή την αρχή τα κράτη-μέλη ε, να χρησιμοποιήσουν και τα ίδια τα δικά τους ε, κονδύλια και τους δικούς τους ανθρώπινους πόρους έτσι ώστε η συνεργασία αυτή να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να προχωρήσει σωστά. Εκτιμούμε το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο σε αυτόν τον τομέα έχει παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο μέσα από διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά projects τα οποία οδήγησαν και σε συντονισμό αλλά και στο γεγονός ε, ότι αυτές οι δομές και οι στρατηγικές έγιναν πιο πολύ διοκτησία των κρατών μελών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχόλια ο εισηγητής. Όχι. Δεν... θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία ήδη είπατε. Περιμένω τις Περιμένω τις τροπολογίες σας, γιατί είπαμε η έκθεσή μου δεν θα έχει σαν στόχο να περιγράψει απλά την κατάσταση, αλλά να κάνει προτάσεις και ενδείξεις που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές, όπως υπόθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αφήσουμε ανοιχτή την δυνατότητα, ιδιαίτερα στο μεγάλο θέμα των επενδύσεων, να δούμε τι νέες πραγματικότητες μακροοικονομικές μπορεί να υπάρξουν. Δεν έχουμε εδώ κάποιο, δεν είμαστε δέσμοι κάποιας λογικής και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια στενότερη σχέση ανάμεσα στις εμπειρίες και τις μακροοικονομικές στρατηγικές συνεργασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωεπιτροπή περιβάλλοντος θα υιοθετήσει τη γνωμοδότησή της στις 28 Σεπτεμβρίου, η Ρέγγι το Νοέμβριο, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, η 13η Σεπτεμβρίου, 5 ε, το απόγευμα. Περνάμε τώρα σε μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον, σχετικά με τον ρόλο των περιφερειών στην εφαρμογή του COP21 για τις κλιματολογικές αλλαγές. Είναι μια έκθεση που αποφασίστηκε από τους συντονιστές και την εμπιστεύτηκαν στην συνάδελφο Άγγελα Βαγίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι έχει υπάρξει μεγάλη συνένεση της ε, διεθνούς ε, επιστημονικής κοινότητας ε, για την υπερθέρμανση. Έχει υπάρξει επίσης και αναγνώριση της ευθύνης την οποία έχει η ανθρωπότητα μέχρι τώρα όλα τα αποτελέσματα αυτής της απαράδεκτης στάσης δυστυχώς τις βιώνουμε σε καθημερινή βάση όχι μόνο αύξηση της συχνότητας ε, βίων ε, κλιματολογικών φαινομένων όπως πρόσφατα στην Καραϊβική αλλά και άλλου είδους συνέπειες. Στο Χιούστον οι συνέπειες ε, των πλημμυρικών φαινομένων οφείλεται εμπολής στο ότι τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με μία μελέτη του Πανεπιστημίου του Τέξας, αστικοποιήθηκαν χιλιάδες περιοχές οι οποίες θα έπρεπε αντίθετα να προστατευθούν γιατί ήταν απαραίτητες για την οικολογική ισορροπία της περιοχής. Αυτό έχει οδηγήσει δυστυχώς σε τεράστιες ζημίες, σε απώλειες ανθρωπίνων ζώων και οι φυσικές καταστροφές, η ξηρασία, οι πλημμύρες, ε, οι κυκλώνες, οι τυφώνες κτλ. θα επιταθούν τα επόμενα χρόνια. Οι κλιματολογικές αλλαγές θα είναι τόσο γρήγορες που οι πληθυσμοί του πλανήτη μας δεν θα έχουν τον απαιτούμενο χρόνο έτσι ώστε να προσαρμοστούν και αυτό είναι κάτι που θα οδηγήσει σε περαιτέρω απώλειες ζωής και επίσης στην καλύτερη περίπτωση σε τεράστιες και απρόβλεπτες μεταναστευτικές αρωές. Το 75% λοιπόν του πληθυσμού προβλέπεται ότι θα επηρεαστεί από τα κλιματολογικά φαινόμενα αυτό φυσικά αντιπροσωπεύει και ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται. Οι συνέπειες λοιπόν των κλιματολογικών αλλαγών είναι ήδη προφανείς και εξαρτώνται βέβαια στην έντασή τους ανάλογα με την περιφέρεια και την περιοχή. Πάντως οι κλιματολογικές αλλαγές σύν της άλλης έχουν και κοινωνικές συνέπειες, επιτείνονται οι κοινωνικές διαφορές λόγω των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Προβλήματα στον τομέα της υγείας, ακατάλληλα τρόφιμα, δυσκολίες στην κινητικότητα κτλ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διεξαγωγής της COP21 στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, 195 χώρες στις 2 Δεκεμβρίου του 2015 υιοθέτησαν την Συμφωνία των Παρισίων για την μείωση της εκπομπής καυσαερίων θερμοκηπίου και της ε, προσαρμογής των μέτρων για την προστασία των οικοσυστημάτων. Την Τετάρτη λοιπόν, ε, τέθη την Τετάρτη ε, Ιανουαρίου του 2016 τέθηκε σε ισχύ έτσι ώστε να πετύχουμε ε, μείωση της αύξησης της θερμοκρασίας η οποία δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα επόμενα 20 χρόνια το 1,5, ε, τον 1,5 βαθμό. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία για τη μείωση των εκπομπών και να υπάρξουν προσαρμογές των παραγωγικών μοντέλων με μείωση ακριβώς των εκπομπών. Οι διάφορες χώρες αναλαμβάνουν την ε, υποχρέωση να μειώσουν λοιπόν ε, τα προβληματικά χαρακτηριστικά των τρόπων παραγωγής τους και να ακολουθηθεί συνεπώς μια γενικότερη διεθνής στρατηγική στον τομέα αυτό. Βέβαια γνωρίζουμε την στάση ε, των Ηνωμένων Πολιτειών που απεσύρθησαν. Είναι η δεύτερη χώρα παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα, 15 100 πίσω από την Κίνα που παράγει το 30% εκπομπών καυσαερίων. Ε, νομίζω λοιπόν ότι οι οικονομικά συμφέροντα γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ έχουν την προτεραιότητα σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και ευημερία και δυστυχώς ε, η κατάσταση θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο να διορθωθεί. Το 2015 σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησαν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών στους στόχους ανάπτυξης για τα επόμενα 15 χρόνια. πολέμηση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών σε σχέση με τους στόχους αυτούς γίνεται αναφορά σε μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν στο εσωτερικό επίσης των πόλεων. Βασικό στόχος, σαν παράδειγμα, κατεπήγοντα μέτρα για την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών, στόχος 7, αηφορία και σύγχρονη δυνατότητα ανάπτυξης για όλους, ε, οι αστικές περιοχές, αστικές συγκεντρώσεις θα πρέπει να είναι αηφόρες οικολογικά, βιώσιμες και ασφαλείς για το σύνολο του πληθυσμού. Επίσης μείωση των εκπομπών, το 3 τέταρτα των εκπομπών παράγονται στις αστικές περιοχές, Αυτά όλα λοιπόν έπρεπε να ενταχθούν στα πλαίσια της COP21 για να σχεδιαστούν οι κατάλληλες πολιτικές για τις πόλεις μας και για τις περιφερειές μας και να είμαστε εμείς σαν Ευρώπη υπόδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε αρκετά ευφυείς έτσι ώστε να προτείνουμε ε, λύσεις. Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν και στην ανάπτυξη και στην βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής με αηφόρο τρόπο και κοινωνικά και οικονομικά. Εφόσον συνεχίσουν να εμένουν οι Ηνωμένε Πολιτείες, αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ κακό για τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά μπορεί όμως και η αντίδραση του πληθυσμού να βοηθήσει στο να αντιστραφεί αυτή η στάση. Στόχος λοιπόν για το 20 είναι η μείωση των καυσαερίων κατά 20% σε σχέση με το 1990 ε, το 20% επίσης ε, της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες και να υπάρξει και αύξηση 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας. Επίσης ε, για το 30 μείωση 30% ε, των καυσαερίων, 30% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 27% βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας για το 2050 από 80 με 95% σε σχέση με το 1990. Αυτή είναι η στόχη λοιπόν τους οποίους έχουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική προσαρμογή στις κλιματολογικές αλλαγές προβλέπει και συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες δεν θα ήθελα να σας καθυστερήσω διαβάζοντάς τις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2008 τη λεγόμενο σύμφωνο των δημάρχων ή των δημοτικών αρχών. Πόλες, πόλεις και ε, περιοχές οι οποίες θέλουν σε εθελοντική βάση να ξεπεράσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εθελοντικά επαναλαμβάνω στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας υπάρξουν, υπήρξαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας. Αναλαμβάνουν οι περιοχές αυτές να πετύχουν τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει εμείς κατά 40% όχι κατά 20% και να υιοθετήσουν επίσης συνολικές πολιτικές για τη μετρίαση των συνεπειών των αρνητικών εννοείται των κλιματολογικών αλλαγών πολιτικών οι οποίες να είναι αηφόρες ε, περιβαλλοντικά. Ε, επίσης ήδη από τις αρχές του 2017 θα τεθεί σε λειτουργία η συμφωνία αυτή των Δήμων για το κλίμα και την ενέργεια οι πόλεις μπορούν να συμμετέχουν ε, όχι μόνο αυτές που είναι ήδη στο εσωτερικό του συμφώνου αυτού αλλά και άλλες να πάρουν μέρος ε, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ήδη από τον προηγούμενο μήνα υπάρχουν 7.000 πόλεις και περιοχές πάνω από 200 εκατομμύρια εκπροσωπούν κατά τη διάρκεια του 2016 στη συνάντηση την ανεπίσημη των υπεύθυνων υπουργών για τις αστικές περιοχές υιοθετήθηκε και η Συμφωνία του Άμστερνταμ για τον καθορισμό της πολιτικής στον τομέα των πόλεων στα πλαίσια μιας νέας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των αστικών περιοχών όπου οι τοπικές αρχές, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι μπορούν να συνεργαστούν. Στα πλαίσια λοιπόν και των στόχων των κοινοτικών πολιτικών, βελτίωση της γνώσης και της εφαρμογής των μέτρων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται βασίζεται και στις εμπειρίες των εταιρικών συμφωνιών που έχουν υπάρξει μέχρι τώρα, συνδεδεμένων άμεσα ή έμεσα με τις πολιτικές που ακολουθούνται στον τομέα των κλιματολογικών, αναζωγόνηση περιοχών, υποδοχή ε, προσφύγων, κυκλική οικονομία, ε, κίνητρα για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, ενεργειακή μετάβαση, αηφόρος ε, πρόταση λύσεων στον τομέα των οικολογικό, κινητικότητα στις αστικές περιοχές, ψηφιακή καινοτομία, η ανάπτυξη όλων αυτών των θεμάτων μπορεί να γίνει στα πλαίσια λοιπόν και των μέτρων τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια της έκθεσής μας λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επιβεβαιώσουμε την σταθερότητα την οποία επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της καταπολέμησης των συνεπειών της κλιματολογικής κρίσης και των κλιματολογικών αλλαγών. Έτσι μόνο θα βρούμε τα κατάλληλα μέτρα, τις κατάλληλες λύσεις για τις ανάγκες των πολιτών μας με αηφορία και εγγυόμενοι ότι οι μελλοντικέ γενιές όχι μόνο θα σώσουν τον πλανήτη και θα τον βρουν στις ίδιες συνθήκες που τον βρήκαμε εμείς, αλλά ακόμα και με βελτιώσεις αν αυτό είναι δυνατόν. Οι πόλεις έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη στα πλαίσια αυτής της συνολικής προσπάθειας, γιατί είναι σημεία θα έλεγα πολύ ευάλωτα και μπορούν όμως να δώσουν λύσεις, να δείξουν λύσεις, έτσι ώστε για να κατανοήσουμε κιόλας ότι τα περισσότερα καυσαέρια ε, παράγονται στις αστικές περιοχές. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν όπως οι τοπικές οργανώσεις, οι πολεοδομικές ρυθμίσεις, η θέρμανση, η, η παραγωγικότητα στον τομέα της αποδοτικότητα, συγγνώμη, στον τομέα της θέρμανσης των κτηρίων, Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των αστικών περιοχών. Θα πρέπει όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε για να βρούμε και τις κατάλληλες ε, πολιτικές. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς οι οποίοι εμπλέκονται και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Όλοι έχουν θεμητό συμφέρον να πάρουν μέρος στην προσπάθεια αυτή έτσι ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. Νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι συντονισμένες σε όλους τους τομείς και αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των λύσεων. Σήμερα είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όλες οι προτάσεις σας θα είναι χρήσιμες και απαραίτητες. Να θυμίσω ότι οι κλιματολογικές αλλαγές δεν έχουν πολιτική ιδεολογία. Η έκθεση αυτή στην ουσία θα αποτελείται από τρία μέρη. Καταρχάς, ε, καθορισμός ενός συγκεκριμένου πλαισίου απαραίτητου για την αποτελεσματική περιγραφή της κατάστασης. Δεύτερον, μια προσπάθεια ορισμού των πολιτικών που θα πρέπει να εφαρμοστούν για τις αστικές περιοχές και τις πόλεις και τρίτον, μια σειρά συστάσεων για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την πολιτική συνοχής. Νομίζω ότι για να μπορέσει κανείς να ορίσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο γύρω από αυτό, είναι απαραίτητο να καθοριστούν ακριβώς αυτά οι εθνικοί και περιφερειακοί στόχοι και στον τομέα της εκποπής αερίων του, του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσης του άνθρακα, αύξηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και μείωση της ενέργειας η οποία καταναλώνεται και επίσης διόρθωση και του συστήματος επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας έτσι ώστε να διατηρήσουμε υψηλή και την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη και να λάβουμε υπόψη μας και την κοινωνική διάσταση. Μια μετάβαση που απαιτεί αλλαγές στον τομέα τον οικονομικό, τον χρηματοδοτικό και τον τεχνολογικό. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια σαφής συνοχή στον τομέα ανάμεσα στις περιβαλλοντικές πολιτικές και στις υπόλοιπες πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν την ισορροπία αυτή σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης είναι απαραίτητη η συμπληρωματικότητα των απαντήσεων στις κλιματολογικές αλλαγές, στη μετρίαση των συνεπειών τους και στην προσαρμογή. <coughs> Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις πραγματικές αιτίες των κλιματολογικών αλλαγών μέσα από τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, της αύξησης της αποδοτικότητας και της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε και τις αρνητικές επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών, να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις ζημίες οι οποίες προκαλούνται σε τομείς όπως η οικοδομή ή μεταφορές, απόβλητα, πολεοδομικές ρυθμίσεις, διαχείριση γενικότερα των πόλεων, και να καθορίσουμε επίσης και τους διάφορους τομείς οι οποίοι θα επηρεαστούν από τις πολιτικές αυτές. Σωστή διακυβέρνηση, συνεργασία, προγραμματισμός, παρακολούθηση των εξελίξεων, συνέχεια των πολιτικών που ακολουθούνται. Έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα μέσα από ένα όραμα θα έλεγα για τις μεγάλες διαφορετικές αλλαγές και στις μεθόδους παραγωγής και στις μεθόδους κατανάλωσης και στις πολιτικές μορφές ε, διαχείρισης ε, των φαινομένων αυτών. Κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η συνειδητοποίηση ε, και η γνώση από πλευράς του πληθυσμού για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, και οι διαφορετικές αλλαγές. Υπάρχει αύξηση επίσης, πρέπει να υπάρχει αύξηση των αρμοδιοτήτων των περιφερειών, έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να προσπαθήσουμε να τα καταστήσουμε αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητη η περιφερειακή συνεργασία και θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε και υπόψη μας και την λογική των φύλων. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με την πολιτική συνοχής δεν μπορεί να, αγνοεί, να αγνοεί τις κλιματολογικές αλές. έτσι ώστε οι πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουν να συνεισφέρουν με συγκεκριμένο τρόπο Κοιτάξτε έχετε ένα λεπτό ακόμα λέει ο πρόεδρος έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους ε, που έχουμε στον τομέα του κλίματος, ε, που είναι εξίσου τουλάχιστον φιλόδοξοι και με τους στόχους της COP21. Στα πλαίσια της συνοχής ε, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα μέτρα από τη μία και τις προσπάθειες διαφοροποίησης με τα μέτρα μετρίασης των αποτελεσμάτων από την άλλη. Νομίζω εδώ έχουμε και ένα παράδειγμα έλλειψης, ε, θα έλεγα, συντονισμού Εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα, αναφέρομαι γενικά στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο όμως να μην αγνοήσουμε συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα για την έλλειψη, κοιτάξτε θα σας σταματήσω λέει ο πρόεδρος, ε, θα σας σταματήσω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε περιορισμένο χρόνο και στη διερμηνία από εδώ και πέρα. Ε, νομίζω ότι καταλάβαμε το πνεύμα της παρέμβασής σας μετά από το σύνορα και μετά από μια πάρα πολύ λεπτομερή παρουσίαση. Καταλάβαμε λοιπόν τι ακριβώς θα λέει η έκθεσή σας η οποία θα μας παρουσιαστεί τον μήνα Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους διάφορους συντονιστές. Η κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να σας πω κάποιες αρχικές σκέψεις για την έκθεση, αν και δεν θεωρώ ότι με μία έκθεση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το μεγάλο θέμα. Θα μιλήσω για το ρόλο των περιφερειών και των πόλεων όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή. Όπως ξέρετε, η COP21 απαιτεί από τις περιφερειακές αρχές να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους επικεντρωθώ στην πολιτική συνοχής γιατί αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και, και σε τρεις θεματικές ενότητες συγκεκριμένα. Στον στόχο 4, ο οποίος είναι η υποστήριξη της οικονομίας προς ε, μια χαμηλή εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, ε, προσαρμογή ε, και η θεματική ενότητα 6 ε, η αποτελεσματικότητα των πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η παρουσίαση που έγινε στην Επιτροπή μας ε, πέρυσι ε, έδειξε ότι 56 δις ευρώ δίνονται για την κλιματική αλλαγή. Αν με ρωτήσετε αν αυτό αρκεί, δεν αρκεί. Σε αυτή την περίπτωση όμως οι χορηγήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Γι' αυτό είμαι πρόθυμη να συζητήσω για τον ρόλο των επιπλέον χρηματοπιστωτικών εργαλείων που θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα project για την κλιματική αλλαγή. Στο ΕΛΚ είμαστε τελείως κατά των δεσμευτικών στόχων, ειδικά για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Τούτου λεχθέντος ε, θέλω να έχουμε συνεργασία με την εισηγήτρια για να μπορεί να, να, να αποφύγουμε τυχόν αλληλοεπικαλύψεις. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ πολύ για τους σοσιαλιστές, ο Ζωζεφ Μοσκό. η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που έχει βεβαίως επιπτώσεις για όλους. Σε διεθνές επίπεδο για την οικονομική ανάπτυξη, για την φτώχεια, για την αύξηση του πληθυσμού και για την έλλειψη των πόρων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να συνεργαστούν όλοι οι δυνατοί τομείς είναι ανάγκη να θέσουμε σε λειτουργία όλες τις πρωτοβουλίες για την βιώσιμη ανάπτυξη. Να υπάρξει διατμηματική συνεργασία, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε μία θέση και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή σε διεθνές επίπεδο. Να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει ποιες ακριβώς είναι οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ούτως ώστε να αλλάξουν τις συνήθειές τους, να αλλάξουν βλαβερές συνήθειες σε ό,τι αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Να υπάρξει μια σημαντική συνδρομή, ούτως ώστε να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη παρόμοια προγράμματα θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους κόσμου, τον κόσμο να καταλάβει ποιες ακριβώς είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Για να το καταφέρουμε πρέπει να ενδυναμώσουμε τις δυνατότητες των διαφόρων κρατών μελών να εκπαιδεύουν τους πολίτες ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Στα σχολεία, για παράδειγμα, να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Θέλω να σας πω, Πρόεδρε, ότι η συνάδελφος Τανσέλα έπρεπε να κάνει την παρέμβαση αυτή. Την έκανα εγώ εκ μέρους της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει να μιλήσει για το Άλντε. Το λόγο έχει ο συνάδελφος από την Ολλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Τις προηγούμενες εβδομάδες παρατηρήσαμε βροχές στην Νοτιοανατολική Ασία και βεβαίως τον τυφώνα στην, αυτή τη στιγμή στην Καραϊβική και στην Αμερική. Παράλληλα στην Αφρική η κλιματική αλλαγή δημιουργεί κλιματικούς πρόσφυγες. Και βεβαίως η ανθρώπινη δράση είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά αυτές τις, αυτά τα, τα φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η συμφωνία του Παρισιού ήταν η πρώτη σημαντική, φιλόδοξη συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν οι δυνατότητες αν μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε ορθά. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αποσυρθεί παρά τα επιστημονικά στοιχεία που παρά τα επιστημονικά στοιχεία που στηρίζουν την ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε και να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία του Παρισιού ό,τι είναι εποφελές σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο είναι εποφελές και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Πρέπει να πείσουμε όλους τους πολίτες όμως σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιφέρειες να αλλάξουν τις συνήθειές τους ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν και αυτοί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τέτοιου τύπου φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, ε, τυφώνες, φαινόμενα τα οποία θα γίνουν όλο και πιο συχνά. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αποφύγουμε ακόμη και αν εφαρμόσουμε τα όσα συμφωνήθηκαν ε, στο Παρίσι. Θέλω να συμπληρώσω τέλος ότι οι προσπάθειες που κάνουμε θα πρέπει να, να καταγράφονται και σε τοπικό επίπεδο των πόλων. Για παράδειγμα, η μετάβαση σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι κάτι που θα πρέπει να καταγράφεται, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε για τους πράσινους τώρα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δύο στους τρεις πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένουν ε, σε πόλεις οι οποίες ε, χρησιμοποιούν το 1 πέμπτο της ενέργειας ε, και δημιουργούν συνεχώς μόλυνση. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Είναι ξεκάθαρο πως οι αποτελεσματικές πολιτικές στην ουσία θα κριθούν από το κατά πόσο μπορούν να εξασφαλίσουν ένα πιο ασφαλές μέλλον. Η στρατηγική COP21 του Παρισιού στην ουσία αναφέρει τα κενά σε αυτό το επίπεδο. Τα κράτη-μέλη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να δώσουν ε, ένα 20% των μακροχρόνιων επενδύσεών τους σε αυτόν τον τομέα. Το 1 τέταρτο των μέσων ε, συνοχής ε, είναι ακριβώς για το θέμα της κλιματολογικής αλλαγής. Τίθεται λοιπόν συνεχώς το ερώτημα κατά πόσον αυτά τα χρηματοδατικά εργαλεία εφαρμόζονται στοχευμένα οι στόχοι έχουν ε, διατυπωθεί ξεκάθαρα. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα διοικητικά μέτρα που θα μπορέσουν να μας επιτρέψουν να υπολογίσουμε αυτά τα εργαλεία χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής αλλά και όλα τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να βοηθούν τα κράτη-μέλη να επιτύχουν τους στόχους ε, της ε, Συμφωνίας του Παρισιού. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα εργαλεία ε, και πώς θα ληφθούν, θα μέτρα σε τοπικό επίπεδο με σκοπό να έχουμε ε, μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, να έχουμε πιο αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση, να δοθούν κίνητρα. Οι περιφέρειες επίσης ε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως το δυναμικό τους. Δεν πρέπει να εφαρμόζουν τις ε, εθνικές γραμμές, αλλά θα πρέπει τοπικά να είναι υπεύθυνε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτό ισχύει για όλους τους τομείς. Τις μεταφορές, την ενέργεια για παράδειγμα, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που έχουν προέλθει, έχουν αντιληφθεί από τη συνεργασία με άλλες περιφέρειες. Και ε, η οποία έχει επιτευχθεί μέσα από χρηματοδότηση, ε, μέσα από προγράμματα. Υπάρχει μια επανάσταση που προϊονίζεται στον τομέα της ενέργειας. Δεν είναι μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να υπάρχει αποκέντρωση των πηγών ενέργειας και η κατανάλωση της ενέργειας ε, θα πρέπει, η ενέργεια θα πρέπει να παράγεται εκεί που καταναλώνεται. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε δίκτυα ενεργειακά σε όλα τα επίπεδα. Η πράσινη ενέργεια είναι αυτή που θα πρέπει κατά πρώτον να είναι διαθέσιμη η βιομηχανία. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να οδηγηθεί σε μια πράσινη μετάβαση, σε μια πράσινη μεταρρύθμιση. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό οι επιστήμονες να βάλουν και αυτοί το λιθαράκι τους. Να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την επιστημονική πρόοδο. Τώρα θα μιλήσω λίγο για τα εξωτερικά στοιχεία. Παρόλο που αυτή η έκθεση αναφέρεται μόνο στις πόλεις, οι πόλεις ε, δεν ε, είναι αυθύπαρκτες. Θα πρέπει επίσης ε, κατά τη μετάβαση από την εποχή των ορυκτών καυσίμων στην νέα εποχή να έχουμε υπόψη μας ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο όσα μας δίνουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σκιώδης εισηγητής δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σάμπερς. Όχι. Η Ρόζα. Η Ρόζα Νταμάτο έχει το λόγο. Grazie Presidente. Eh, il tema Ευχαριστώ. Η έκθεση για το COP21 και την πολιτική συνοχή έχει πολύ μεγάλη σημασία για το κίνημα των πέντε αστέρων. Ελπίζουμε από την κυρία Βαλίνα λοιπόν αρκετές προτάσεις. Όπως λέγαμε ήδη το Δεκέμβριο του 2015 δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από τη Συμφωνία των Παρισίων συνειδητοποιούμε ότι οι αλλαγές θα πρέπει να λάβουν υπόψη την πραγματική οικονομία και δεν μπορεί να υπάρξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με επιλογές θαραλέες και δραστικές. Απλά μειώνουμε τις ζημίες αν θέλετε. Στην ουσία μένουμε κάτω από την αύξηση ε, των δύο ε, βαθμών, γύρω στο 1,5 και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τα σωστά γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε όπως πάμε τώρα θα αυξήσουμε για δύο βαθμούς την θερμοκρασία του πλανήτη. Σύμφωνα και με τις, ε, την τεκμηρίωση από πλευράς ε, των Ηνωμένων Εθνών βλέπουμε ότι κάποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ε, άμεσα τα μέτρα για να αποφύγουμε την αύξηση πάνω από το 1,5%. Ε, πάνω από το 80% των τελικών φυσικών καταστροφών οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα τα οποία συνδέονται θα έλεγα με ακραίες μετεωρολογικές εκδηλώσεις οδήγησαν σε 607.000 απώλειες, μάλλον 607.000 ανθρώπινων ζωών στον κόσμο όλο. Το 15 αυτά, το 16 τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε μέσω της πολιτικής συνοχής για να βοηθήσουμε. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξουμε μια πραγματική πολιτική απεμπλοκής από τον άνθρακα και με μαζικές επενδύσεις στην περιφερειακές πολιτικές. Υπάρχουν χώρες οι οποίες αποφάσισαν να φύγουν ε, από την COP21 και τις καταδικάζουμε. Αλλά τι θέλουμε εμείς σε σχέση με την Ευρώπη. Ναι, η Ευρώπη μέσω του ΕΦΣΥ, του Στρατηγικού Ταμείου, χρηματοδοτεί τον άνθρακα. Οι θάλασσές μας, ιδιαίτερα η Αδριατική, ε, ε, και, το Ιόνιο πέλαγος ε, μαστίζονται από, αυξημένα ακραία οικολογικά φαινόμενα. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Οι αλλαγές θα πρέπει να ξεκινήσουν από εμά τους ίδιους. La riduzione concreta delle emissioni come un elemento chiave di valutazione della Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε στη λογική αυτών των λειτουργικών προγραμμάτων και να μην έχουμε παρά μια στρατηγική συνεκτική μακροπρόθεσμα να στοχεύει στην απομάκρυνση από τον άνθρακα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τον άνθρακα, αλλά όλες τις ορυκτές πηγές ενέργειας, μεταξύ των οποίων και το φυσικό αέριο πρέπει να προωθήσουμε μια στρατηγική θα έλεγα η οποία ανακαλύπτει και τα δίκτυα μεταφοράς και εγκατέλειψης των ορυκτών καυσίμων. Πρέπει εμείς λοιπόν να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις για την πολιτική μετά το 2020 πριν είναι αργά. Ευχαριστώ, θα ήταν λάθος μου να μην σας ακούσω. Ευχαριστώ και τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο που και τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα. Ε, θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ρέγγιο. Συνεννοηθείτε ποιος θέλει το λόγο. Διαφορετικός εκπρόσωπος, διαφορετική γενική διεύθυνση, εκπροσωπούμε το ίδιο όργανο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Θα μιλήσω αγγλικά τώρα. Πίστευω ότι ολόκληρος ο κόσμος μπορεί να στηρίζεται στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στα επόμενα χρόνια είναι να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες μας, να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι παρούσα την επόμενη εβδομάδα στο Μοντρεάλ, από κοινού μαζί με την Κίνα και τον Καναδά, αλλά και άλλες χώρες, ακριβώς για να ενδυναμώσουμε τις συμμαχίες μας ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Όπως ήδη υπόθηκε, η κλιματική αλλαγή τόσο σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση όσο και την προσαρμογή είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο. Και η Συμφωνία του Παρισίου για πρώτη φορά αναγνώρισε το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων, των χωρών, ούτω ώστε να μπορέσουμε να περικόψουμε τις εκπομπές βλαβερών αερίων, να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητά μας αλλά και να προωθήσουμε τη συνεργασία μας. Υπάρχουν πάντοτε δύο όψεις σε κάθε νόμισμα. Οπότε, ναι, οι πόλεις αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, το έχουμε όλοι παρατηρήσει μέσω των διαφόρων καυσώνων που αντιμετωπίζουμε. Ε, εμένα προσωπικά μου έχουν κινήσει το ενδιαφέρον αρκετές πόλεις και χώρες όπου το έχουν ε, αναδείξει σε επιχείρηση το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που κάνουμε λοιπόν στο τοπικό επίπεδο είναι να στηρίζουμε την τοπική ευθοδιοίκηση και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν 7.500 πόλεις σήμερα που συμμετέχουν στο δίκτυό μας και έχουν υιοθετήσει στρατηγικές προσαρμογής. Εθνικά έχουμε 24, με έχουμε 24 κράτη-μέλη τα οποία έχουν τέτοιου τύπου σχέδια προσαρμογής. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο όλα τα στοιχεία αυτά που σας αναφέρω είναι α, διαθέσιμα βέβαια στο διαδίκτυο, αλλά και προσωπικά μπορώ να σας τα παραδώσω αν τα χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δράση των δικτύων των δημαρχείων, πρόκειται για δεσμεύσεις, πρόκειται για τοπικές συμβολές, γιατί κάθε χρήση, κάθε, με συγχωρείτε, περιοχή αποφασίζει με ποιο τρόπο θέλει να συνεισφέρει. Για το 2020 η σύνοδος των δημάρχων έχουν ήδη καταφέρει το 23% των όσων έχουν δεσμευτεί να κάνουν. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Αναφέρθηκε ήδη ότι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σύνοδο των Δημάρχων έχει οδηγήσει σε μια σύνοδο η οποία ονομάζεται Παγκόσμια Σύνοδος Δημάρχων. Είναι η αντιπροσωπεία μας στην Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Θα συναντηθούν για την COP23, θα ανταλλάξουν στοιχεία σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές. Το 2018 η... τα Ηνωμένα Έθνη θα προωθήσουν το διάλογο μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών και τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε να δουν πώς αυτή η συλλογική προσπάθεια μπορεί να βοηθήσει. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην έκτη έκθεση εκτίμησης σε ό,τι αφορά τις διάφορες πόλεις δεν έχουμε ακόμη το χρονοδιάγραμμα για την έβδομη τοπική δράση να στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής και να εφαρμόζει τα όσα καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Και θέλω να πω σε όλους σας που δεν έχετε συμμετάσχει σε αυτή την ε, Δημαρχιακή Σύνοδο να α, αναλάβετε δράσεις, όποια πόλη και αν βρίσκεστε. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, θα πρέπει να σας σταματήσω. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, αν μπορείτε απλά να φτάσετε στο συμπέρασμα. Απλά να σας πω, λέει η ομιλήτρια, σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων έχουμε αυτά που είναι ταμεία αρρωγής να βοηθήσουν στην οργάνωση των επενδύσεων. Έναντι συμπεράσματος σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή σήμερα και μετά όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένε Πολιτείε, οι τοπικοί φορείς έχουν ένα σημαντικό ρόλο να, διαπραγμα... να, δια... να παίξουν και η πρόκληση μπροστά μας είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας τρομάξει, αλλά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα υπάρξει α, και άλλη παρουσίαση το Νοέμβριο η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα πλούσια. Ευχαριστώ θερμά την ε, συναδελφό μας Βελίνα για την ενδελεχή παρουσίασή της. Σε ό,τι αφορά την σημασία του πόσο πρέπει να συμμετάσχουν οι τοπικοί φορείς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα όσα συμφωνήσαμε στην COP21. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Κλείνω την συνεδρίαση αυτή. Όσοι συμμετέσχουν στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών μπορούν να παραμείνουν. να σας υπενθυμίσω τις δύο συναντήσεις σήμερα το απόγευμα. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι έχουν πολλά να ρωτήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ σε όλους, ευχαριστώ όλους και ευχαριστούμε πολύ και την Επιτροπή.